Good morning, dear colleagues. Sorry for the slight delay. Um, it was unexpected. Καλημέρα συνάδελφοι, μικρή καθυστέρηση. Συγχωρέστε μας γιατί αντικαθιστώ την κυρία Βαλεάν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το πρώτο θέμα είναι η έκρηση της ημερήσιας διάταξης. Και αν δεν υπάρχει... Α, συγγνώμη το σημείο 8 του σχεδίου γνωμοδότησης για την ανανεώσιμες να αλλάξει θέση με το σημείο 9 της κυρίας Γκροστέτ για την αναλογικότητα για τα νέα επαγγέλματα. Δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις για την αλλαγή της σειράς αυτή. Και αν συμφωνούν και οι δύο εισηγητές, μπορεί έτσι να εγκριθεί τροποποιημένη ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω κανέναν να ενίσταται. Ωραία. Αγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Ανημερωτικά να σας πω ότι για την τερμηνία έχουμε τερμηνία σε 20 γλώσσες. Εστονικά, λατωνικά, μαλτέζικα και εγώ αδελικά δεν έχουμε. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους που θα θέλανε να παρακολουθήσουν στη μητρική τους γλώσσα και δεν μπορούν. Και έχετε στην ε, εφαρμογή e-meeting τα έγγραφα της συνεδρίασης και η συνεδρίασή μας όπως πάντα δημοσιεύεται στο διαδικτύο. Στο σημείο 3. Ανακοινώσει σε ό,τι αφορά τις συστάσεις των συντονιστών για τις 21 Ιουνίου 2017. Οι συστάσεις των συντονιστών σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Να ζητήσω από τους συναδέλφους αν έχουν αντιρρήσεις. Όχι. Εγκρίνονται λοιπόν οι συστάσεις. Στο σημείο 4 πάλι τα πρακτικά της συνεδρίασης της 24 Απριλίου 2017 και 25 Απριλίου έχουμε να εγκρίνουμε. Αν δεν λάβουμε καμία παρατηρήση μέχρι το τέλος της συνεδρίαση θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Και ας περάσουμε στο σημείο 6. Το σημείο 5 θα μας το παρουσιάσει η πρόεδρος μόλις καταφτάσει. Και έτσι λοιπόν περνάμε στο σημείο 6. Έκθεση Φάρια. διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μα στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030. Και θα ήθελα να δώσω καταρχά το λόγο στον κύριο Χωσέ Ινάσιο Φαρία. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Και θα ήθελα να καλωσορίσω Κάποιου καλεσμένου που έχουμε μαζί μας, ο κύριο Σίμετς από το ε, Συμβούλιο και από την ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Υπό την ιδιότητά μου ως εισηγητής για το θέμα αυτό με τον μακροσκελή αυτό τίτλο που έχει να κάνει με την ατζέντα για το 2030 και τους ε, στόχους βίωσιμης ανάπτυξης να ευχαριστήσω την, την Επιτροπή Μεταφορών καταρχάς για την γνωμοδότησή της. Η κυρία Μούντερ Ντραγκιά είναι η εισηγητρία και θα ήθελα να καλωσορίσω και τον κύριο Σάιμοντς, ο οποίος είναι εισηγητής από την ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για το θέμα αυτό και ο οποίος μας παρουσίασε τη δική του αντίληψη και τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Η κοινή ανακοίνωση για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης των θάλασσών. Ιδιαίτερα όπως ορίζεται στην, στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα να λάβει ηγετικό ρόλο για την ενίσχυση τη Διεθνού Διακυβέρνηση των ωκεανών ω τμήμα συντονισμένων προσπαθειών που γίνονται από πλευρά της διεθνού κοινότητα. και η ατζέντα για το 2030 εντόπισε τα μέτρα αυτά για τις θάλασσες ως ε, ένα από τα 17 απαραίτητα μέτρα για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το σημείο υπερθμών 14 για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Τα διεθνή λοιπόν σώματα αντιλαμβάνονται τη σημασία της τη βιώσιμη ε, αξιοποίηση των ωκεανών προκειμένου να διατηρηθεί και η βιοποικιλότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Και αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη της ατζέντα του 2030. Οι ωκεανοί και τα θαλάσσια, οι θαλάσσιοι πόροι είναι ουσιώδους σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη και την οικονομική ανάπτυξη και για όλο μα τον πλανήτη. Η διασυνοριακή δε ε, φύση της διαχείρισης των ωκεανών προαπαιτεί συνεργασία μεταξύ των κρατών προκειμένου να καταφέρουμε να διαχειριστούμε το θέμα των θαλασσών με πραγματικά βιώσιμο τρόπο. Και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, σοβαρά προβλήματα που αποτυπώνουν την υγεία, αν θέλετε, των θαλασσών που βρίσκεται υπό απειλή απειλείται με μη αναστρέψιμες ζημιές λόγω της αλλαγής του κλίματος και αυτό είναι ήδη σαφές και ορατό σε διάφορες περιστάσεις. Για πρώτη φορά λοιπόν ε, είναι σαφής η σύνδεση μεταξύ της αλλαγής του κλίματος και των ωκεανών και των θαλασσών. Νομίζω ότι πρόκειται για ιστορικό επίτευγμα, το υπογραμμίζουμε. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει διάφορα σημεία σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη διαχείριση των θαλασσών και κατά δεύτερον άσκηση πίεση σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική ενίσχυση των θαλασσών, το θέμα των θαλασσών μεταφορών και κατά τέταρτον η δημιουργία ενός πλαισίου για πιο στενερά στοιχεία και έρευνα σε ό,τι αφορά τις θάλασσες. Οι θάλασσες λοιπόν πλήττονται από τον αντίκτυπο του διοξιδίου του άνθρακα. Και τα θαλάσσια οικοσυστήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικέ λύσει. Επίση, μα απασχολούν ιδιαίτερα το θέμα των λιμάτων στου ωκεανού και στι θάλασσε. Αυτό αφορά όλε τι περιοχέ του πλανήτη. Θα πρέπει να αναπτύξουμε λοιπόν και ατομικέ λύσει. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ε, γνώση και την ευαισθητοποίηση για τι θάλασσε και να υπογραμμίσουμε τη σημασία τη βιώσιμη θαλάσσια οικονομία, τη μπλε οικονομίας, όπως ονομάζεται. Και αυτό προφανώς αποτελεί ένα τμήμα της γενικότερης προσέγγισης μας για τη βελτίωση των όρων και των συνθήκων για τις πριν από το 2020 σε ό,τι αφορά επίσης την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά πλαστικά και για άλλα λίμματα στις θάλασσες. Μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν όλα τα στοιχεία αυτά, όλα τα προβλήματα αυτά, χρειάζεται καλύτερη διεθνή διακυβέρνηση και με τον τρόπο αυτό θα είναι πιο εύκολη και η υλοποίηση τη περιφερειακή συνεργασία Οι εταιρικέ σχέσεις με του βασικού ε, εμπλεκόμενου φορεί θα πρέπει να ενισχυθεί ω τμήμα τη γενικότερη, διεθνού διακυβέρνηση των θαλασσών. Και νομίζω ότι αυτέ οι σχέσεις συνεργασία οι εταιρικέ σχέσει είναι το κλειδί εδώ για να πετύχουμε καλύτερη διακυβέρνηση των ωκεανών και διαχείριση των ωκεανών. Να ευχαριστήσω κλείνοντα όλου του συναδέλφου που συμμετείχαν στην κατάρτιση του κειμένου αυτού και να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Περιβάλλοντο και το προσωπικό του υπαλλήλου και τη γραμματεία. Προσβλέπω στι παρατηρήσει σα και στα σχόλιά σα, τα οποία είμαι βέβαιο ότι και θα εμπλουτίσουν την έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you. Um, and now I give the floor to the uh, uh, first from the σας ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο στους κυριώδες εισηγητές. Πρώτα απ' όλα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Βόλκαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και τον συνάδελφο Φαρία. σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχέδιο νομοθέτηση αυτό, το σχέδιο έκθεση αυτό, το οποίο καλωσορίζω από πολλέ απόψει και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παραπομπή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση τη βιώσιμη διαχείριση των ωκεανών. Αλλά θα ήθελα να βαθύνω σε ορισμένα σημεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο θα φιλοξενήσει σχετικό, σχετική διάσκεψη στη Μάλτα. Και διαβάζουμε λοιπόν σε ό,τι αφορά την εκδήλωση αυτή στα αγγλικά. Η ανθρωπινή δράση έχει επηρεάσει σοβαρά ρήπανση στους ωκεανού μας ε, μέσω τη εκμετάλλευση, της υποτίμησης και της παγκόσμια ε, θέρμανσης. Και αυτό ε, έχει σοβαρές συνέπειες για όλους. Χρειάζεται ένα νέο όραμα και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ε, με όλα αυτά δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο όραμα και ένα δεσμευτικό στενερό σχέδιο δράση. Ε, σε αυτό θεωρώ ότι συγκαταλείεται και ένα ε, σοβαρό σχέδιο για την παγκόσμια διαχείριση των ωκεανών. Εκεί επικεντρώνεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι άλλε δύο προτεραιότητε με φυσικό σύμφωνο. Η προτεραιότητα για την διεθνή έρευνα για τους ωκεανούς και το πώς μπορούμε να μειώσουμε και να ελαττώσουμε τις πιέσεις που δέχονται οι ωκεανοί και οι θάλασσες. Σε ό,τι αφορά το κατεπήγον του ζητήματο των περιβαλλοντικών ζητημάτων, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπογραμμιστούν λίγο πιο έντονα. Εδώ θέλω να πω ότι πρέπει να εστιαστούμε λίγο παραπάνω, αν θέλουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσουμε να είμαστε ηγετική δύναμη στην προστασία των ωκεανών. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο πολύ το θέμα της προστασίας των ωκεανών, να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι να κάνω προστάσει συμπληρωματικέ σε τέσσερι τομείς. Καταρχά. σε ό,τι αφορά την εκπομπή ε, λιμάτων στην αυτιλία, θα πρέπει να τα ρυθμίσουμε καλύτερα τα πράγματα. Στο Αμβούργο, κοντά, από, κοντά στην πατήδρα μου, η εκπομπή αζότου από τα πλοία είναι πιο μεγάλη από, ότι, από, τα, από τα οχήματα, από τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι μεγάλο κίνδυνο για την υγεία των ε, πολιτών και το 2020 αναφέρεται ότι τα αυτοκίνητα εκπέμπουν πιο πολλά οξύδια ζώτου και αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Οι χώρε, οι πόλει που έχουν μεγάλους λιμένες αναφέρουν ότι λόγω ανταγωνισμού δεν μπορούν να δράσουν ιδιαίτερα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευρωπαϊκή ρύθμιση και θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τα πλοία τα οποία βρίσκονται στους λιμένες να χρησιμοποιούν, να χρησιμοποιούν ηλεκτρικό και να μην χρειάζεται να λειτουργούν και να καίνουν καύσιμα όσο είναι μέσα στο λιμάνι για την εκφόρτωση. Επίσης, χρειαζόμαστε περαιτέρω μέτρα για να μειωθούν οι εκπομπές οξυδίου του αζότου μέσω τεχνικής αναπροσαρμογής του υφιστάμενου στόλου, γιατί είναι τεράστιος και ο κίνδυνος για την υγεία που συνεπάγονται τα οξύδια αζότου. Σε ό,τι αφορά το αζότο, λοιπόν, και άλλες επιδημίες ουσίες, θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, για παράδειγμα, τα όρια ε, στη Μεσόγειο από το 2020 και μετά μπορεί να είναι πενταπλάσια από αυτά που ισχύουν στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα. Χρειαζόμαστε και πιο πολύ έρευνα στον τομέα αυτό. Δεύτερο σημείο τώρα. Όταν, ε, άμα θέλουμε να ενισχύσουμε την διεθνή θα πρέπει να αυξηθεί και η λογοδοσία και η οργάνωση της διεθνούς διαχείρισης. Το σχέδιο του 2018 για τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου θα πρέπει να την εξετάσουμε με επικριτικό πνεύμα, γιατί θεωρούμε ότι μας δίνει υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα και θα πρέπει επίσης να υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των κρατών μελών στους διεθνείς οργανισμούς. Και δεν μπορεί και η ΜΚΟ του τομέα να μην ενημερώνονται και να μην ενημερώνουν για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά το τρίτο σημείο μου τώρα, μπλε ανάπτυξη, αναφέρθηκε αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό εις ε, βάρος ε, του περιβάλλοντος όπου ο κίνδυνος για τη χρήση των φυσικών πόρων είναι ε, υπερβολικά υψηλός, η αρχή της πρόληψης μας υποχρεώνει καταρχάς να προστατεύσουμε τα φυσικά, τα περιβαλλοντικά συστήματα και όχι την οικονομία. Αυτό επίσης σημαίνει, όπως αναφέρεται στην έκθεση, ότι θα πρέπει να ζητήσουμε σχετική, ε, σχετικό προσανατολισμό. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί καλύτερα τους πόρους της. Το τέταρτο και τελευταίο σημείο, η θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται όλο και πιο πολύ χωματερή του πλανήτη. Πλαστικές σακούλες, καλλιντικά, λιπαντικά, όλα αυτά καταλήγουν λίγο πολύ στη θάλασσα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας των θαλασσών και να βοηθήσουν όλες, όλοι οι πολιτικοί κλάδοι. Θα πρέπει μακροπρόθεσμα να αντικατασταθούν 100% τα πλαστικά προϊόντα, να βελτιωθεί η κυκλική οικονομία και να προσέξουμε προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση από τα αφρίτα προστατευτικά. Και άλλο ένα παράδειγμα από την ε, πατρίδα μου, που προστατεύεται από την UNESCO ε, είναι σαφές, ε, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητέ γιατί θεωρώ ότι το, η έκθεση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να βελτιωθούν απλά κάποια σημεία. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές. Είχα ξεχάσει να βάλω κάποιο όριο στο χρόνο γόρευση του πρώτου σκιώδη, επομένω δεν θα μπορούσα να βάλω στου υπόλοιπου. Παρ' όλα αυτά θα σα ζητήσω, εάν μπορείτε, να μην μακρηγορείτε. Επόμενο ομιλητή από την Άλτε, κυρία Μέσνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον ε, Χωσέ Ινάσιο Φαρία. Είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση και εγώ το αντιλαμβάνομαι έτσι. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε ο συγητή και συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε ο συνάδελφο πριν από λίγο. Είναι θετικό το γεγονό ότι στο Ιωβιλέο, αν θέλετε, τη ευρωπαϊκή πολιτική τη θάλασσα που ξεκίνησε το 2007, κοιτάμε και πάλι την πολιτική αυτή. Γιατί η συνολική πολιτική για τις θάλασσες και του ωκεανού δηλώνει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν οι ικανότητε και οι ευκαιρίε που μας προσφέρουν οι θάλασσες, αλλά με βιώσιμο, ισορροπημένο τρόπο. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με ισορροπημένο τρόπο και με μεγάλη προσοχή για να μην γίνει κανένα λάθος. Και αυτό θεωρώ ότι αναπτύσσεται σωστά ω ιδέα με την μπλε αυτή ανάπτυξη, πολύ σωστή ιδέα. Και ξέρουμε ότι οι ωκεανοί είναι απαραίτητοι για την ε, ανθρωπότητα. Μιλάμε για τον μπλε πλανήτη ο ωκεανός χρειάζεται ω πόρος και όχι μόνο για το κλίμα και για το κλίμα ασφαλώς αλλά και για άλλους πόρου, για πρώτες ύλε, για μπλε βιοτεχνολογία, για την ενέργεια όλα αυτά εξαρτώνται και είναι σε στενή συνάρτηση με τους ωκεανούς και φυσικά θα πρέπει να είναι υγιείς οι ωκεανοί που δεν είναι στην παρούσα φάση. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν για να είναι υγιεινοί υγιείς ή ωκεανοί και να μπορούμε λοιπόν να τους αξιοποιήσουμε. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η νέα εκμετάλλευση και αξιοποίηση, να το κοιτάξουμε με επιστημονικό τρόπο για να μην καταρρεύσει το σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή και έχουμε ήδη εργαλεία. Έχουμε τον κανονισμό για τη θαλάσσια τάξη, με τον θαλάσσιο χώρο, συγγνώμη, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο και θέλουμε να επικρατήσει και σε διεθνέ επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορεί να πετύχουμε σε, σε διεθνέ επίπεδο. Η Ευρώπη βρίσκεται σε καλό σημείο σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τι θάλασσε, αλλά θα πρέπει να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο προκειμένου βιώσιμα να προωθήσουμε την αξιοποίηση των ωκεανών. Η ΕΠΑ έχουν παρουσιάσει κάποια ελλείμματα τώρα με τον Πρόεδρο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε και το καλύτερο. Έχουμε πολλούς διεθνείς οργανώσεις ε, τον ΟΗΕ, τον Διεθνή Οργανισμό για τις Θάλασσες και το καθεξής και επίσης έγινε πρόσφατα και τον Ιούνιο μια μεγάλη συνεδρίαση παγκόσμια για τις θάλασσες και τον Οκτώβριο θα λάβει χώρα και στη Μάλτα σχετική εκδήλωση και συνέδριο και προφανώς η στρατηγική για το πλαστικό είναι πολύ σημαντική. Σε ό,τι λοιπόν τα πλαστικά, να πω δύο λόγια. Χθες Μόλις διάβασα ένα άρθρο που αναφέρει ότι κάθε λεπτό στον κόσμο αγοράζονται ένα εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια και αυτό θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και αυτό όχι μόνο σε εμά στην Ευρώπη αλλά και στην Ασία όπου επειδή είναι τη μόδα και επειδή υπάρχει και κίνδυνος με το νερό τη βρύση, ε, θα αυξηθεί ακόμα περαιτέρω αυτή η κατανάλωση. Μόνο 7% των ε, μπουκαλιών αυτών δε καταλήγουν στην ανακύκλωση. Και η ανακύκλωση, ξέρετε, ε, εξοικονομεί 75% ενέργεια σε σχέση με την παραγωγή νέων ε, μπουκαλιών. Παρ' όλα αυτά δεν προτιμάται. 6,6% των παραγωγών χρησιμοποιούν, ε, προβαίνουν μάλλον σε ανακύκλωση. Η Coca-Cola είπε για παράδειγμα ότι σκοπεύει να κάνει αλλαγή του εξοπλισμού της και στις χώρες όπου προμηθεύουν τα προϊόντα τους να επιτρέψουν τη χρήση ανακυκλωμένων μπουκαλιών. Είναι πρώτο βήμα, αλλά δεν αρκεί σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε το εξή. Καταρχάς να έχουμε υπόψη ότι 80% των πλαστικών φτάνουν στις θάλασσες μέσω της ε, ξηράς, το είπε και ο Τίμο, και τα πλαστικά αυτά, ναι, ναι, ναι, θα κλείσω πρόεδρε τώρα σε λίγο, αποτελούν ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Για παράδειγμα, από τους G7 ε, προετοιμάζονται σχετική διακήρυξη για τα πλαστικά και έχουμε μια ομάδα από διάφορες πολιτικές ομάδες, μια ομάδα εργασία για τα πλαστικά. Σε αυτή την ομάδα λοιπόν με τους συναδέλφους προσπαθούμε να τοποθετηθούμε σε ό,τι αφορά τη μελλοντική στάση του Κοινοβουλίου προκειμένου να αντιληφθούν όλοι πιο πολύ την, το καταπίτωτο χαρακτήρα. Τελευταίο, τελευταίο σημείο για τον ε, ορίζοντα 2020. Χρειαζόμαστε μέσα προκειμένου να υπάρχει σωστή α, προώθηση των θεμάτων των επιστημονικών αναφορικά με τους ωκεανούς και τις βαθιές θάλασσες. Ευχαριστώ. Ο επόμενος από την, ε, από την euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για την υψηλή ποιότητα έκθεση που μας παρουσιάζει. Γνωρίζετε ότι προέρχομαι από μια εκλογική περιφέρεια η οποία είναι πλέον απομακρυσμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πλέον ναυτική. Πρόκειται για μια εκλογική περιφέρεια η οποία καλύπτει ωκεανούς και συνολικά καλύπτει 11 εκατομμύρια ε, τετραγωνικά χιλιόμετρα ε, των υπερπόντιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, της, της Γαλλίας. Και, ε, πιστεύω ότι οι χώρες αυτές που βρίσκονται στην Καραϊβική, στον Ινδικό ωκεανό, στον Ειρηνικό ωκεανό, είναι χώρες οι οποίες στη μεγάλη τους πλειονότητα υπήρξαν απικίες. Και γνωρίζουμε ότι στη διάρκεια της ιστορίας η θάλασσα, η, ο έλεγχος των θαλασσών και των ωκεανών ήταν ένας από, τους, από τα βασικά κίνητρα που οδήγησαν στις, ε, στην απεικιοκρατία. Και για την α, ένα άλλο κίνητρο ήταν προφανώς η χρήση των φυσικών πόρων αυτών των περιοχών. Ανησυχούμε λοιπόν όταν διαπιστώνουμε ότι οι παλές απεικιοκρατικές δυνάμεις ε, είναι, συνεχίζουν να είναι έτοιμες να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους των χωρών μας. Γι' αυτό και από αυτό το πρίσμα βλέπουμε τη σημασία της διεθνούς διακυβέρνησης της χρήσης των ωκεανών, της προστασίας των ωκεανών. Είναι ένα θέμα τεράστιας σημασίας για ολόκληρη την ανθρωπότητα για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούμε την ε, αλλαγή του κλίματος, την υπερθέρμανση του πλανήτη και αυτό που καθιστά το, θέμα ακόμα πιο σοβαρό και δύσκολο σήμερα είναι ότι έχουν συνδυαστεί μια σειρά παράγοντες ε, που επιβαρύνουν τους ωκεανούς, ορισμένοι αναφέρθηκαν. Πρώτον η δημογραφική αύξηση, και η πίεση στο φυσικό περιβάλλον που αυτή δημιουργεί είναι η κλιματική αλλαγή και αυτό που αναφέρεται ως και η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων των ωκεανών. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν καλούμαστε να δράσουμε. σε αυτές τις περιοχές. Εμείς ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το, ένα, το έκτο κύμα α, εξάλληψης ειδών. Και μας λένε οι επιστήμονες ότι αν συνεχίσουμε με τους σημερινούς ρυθμούς ε, αλίας μέχρι το 2050 δεν θα υπάρχουν πια αλλιεύματα. Για, να λοιπόν ποια είναι και, και γιατί είναι τόσο μεγάλη σημασία η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θα έπρεπε να ε, κοιτάμε πώς να δημιουργήσουμε ένα διεθνές δίκαιο που να ρυθμίζει αυτή τη χρήση των ωκεανών και δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά από αυτό ακόμα. Γνωρίζουμε ότι αυτές δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν να καταβροχθήσουν τους φυσικούς πόρους των ωκεανών δεν θα σταματήσουν αν δεν κάνουμε εμείς κάτι και, για να τις σταματήσουμε. Και ε, σε αυτό πιστεύω ότι εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε να παίξουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Συχνά μιλούμε για τον κατακαιρματισμό που υπάρχει στη διαχείριση των ωκεανών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πράγματι ισχύει αυτό. Και Γι' αυτό χρειάζεται να αλλάξει, να ανανεωθεί το διεθνές πλαίσιο. Σήμερα ψιζόμαστε σε μια συνθήκη του 1982. Χρειάζεται αναθεώρησή της για να επικυρωποιηθεί, για να γίνει πιο συνεκτική και να υπάρξει και μεγαλύτερη διαφάνεια. Συνολικά θα έλεγα ότι υποστηρίζουμε την έκθεση του συναδέλφου. Θα βάλουμε βέβαια και κάποιες προτάσεις. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κλείνουμε το κύκλο συζήτησης με τους... Όχι, κάποιον ξέχασα. Το συγγνώμη. Δεν σας είχα δει κυρία Έγκστρομ από τους πράσινους. Έχετε το λόγο. Μιλάω λοιπόν εξ ονόματος των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ. Καλωσορίσαμε την ανακοίνωση της Επιτροπής για την διακυβέρνηση της διαχείρισης των ωκεανών, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα και πιστεύω ότι η έκθεση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, Θα είχαμε να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε όμως κάποια ερωτήματα προς την Επιτροπή. Τι κάναμε, ε, μάλλον κάναμε κάποια βήματα για να μειωθεί η χρήση των πλαστικών σοκουλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης για την απαγόρευση ε, πλαστικών τα οποία είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον. Όμως αυτές οι πρωτοβουλίες δεν επιλύουν το πρόβλημα άλλων αντικειμένων που είναι φτιαγμένα από πλαστικό και τα οποία, κατα... καταλήγουν στους ωκεανούς. Ιδιαίτερα σήμερα όταν έχουμε ένα σωρό προϊόντα τα οποία έχουν πλαστικές συσκευασίες που έχουν σχεδιαστεί μόνο για να χρησιμοποιούνται λίγα λεπτά και μετά απαιτιώνται. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ε, Πίσω την Επιτροπή τι κάνουμε σε αυτόν τον τομέα, δεδομένου μάλιστα ότι η καταπολέμηση της χρήσης του πλαστικού, η μείωση μάλλον της χρήσης του πλαστικού, ήταν μια από τις ε, σημαντικές πρωτοβουλίες που είχαν αναφερθεί στην προσπάθεια να πάμε προς μια πράσινη οικονομία. Ποιες πρωτοβουλίες λοιπόν προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή σε αυτό το τομέα, γιατί μέχρι στιγμής τα εθελοντικού χαρακτήρα μέτρα δεν έχουν δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή αυτή τη στιγμή προετοιμάζει μια στρατηγική για, τα για το πλαστικό. Έχει ξεκινήσει μια... Μάλλον μόλις τώρα ξεκινάει η διαδικασία διαβούλευσης για τη στρατηγική αυτή. Και το ερώτημά μου είναι πώς θα ήταν δυνατόν αυτό τα συμπεράσματα της διαβούλευσης να ληφθούν υπόψη όταν, έχουμε ήδη, όταν έχει ήδη ξεκινήσει να καταγράφεται, να, εγγράφεται, ή να συγγράφεται μάλλον στρατηγική από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Επίσης υπάρχει το ζήτημα της αλίας στις, στις ανοιχτές, ανοιχτή θάλασσα. Γιατί, συγγνώμη, την εξόριξη ορυκτών καυσίμων στην ανοιχτή θάλασσα. Γιατί προωθείται αυτήν τη ε, πρωτοβουλία όταν γνωρίζουμε την κίνδυνο για το περιβάλλον που, που Και πώς θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις όταν ε, ξεκινούν πρωτοβουλίες αξιοποίησης φυσικών πόρων που βρίσκονται στο, στην υποθελά, στο, στο, βυθό. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διεθνή ύδατα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις περιοχές χρειάζεται μια προστασία σε διεθνές επίπεδο. Όμως, οι διεθνείς οργανισμοί που λειτουργούν για αυτή την κατεύθυνση δεν, λειτουργούν αποτελεσματικά. Και ρωτώ, γιατί δεν έχει κάνει κάποιες προτάσεις για να αναλάβουμε δράση, για να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας του Διεθνούς Οργανισμού Διαχείρισης των Βυθών. Επίση, όσον αφορά τώρα τις σχέσεις με ορισμένα κράτη-μέλη, ορισμένα μέλη του Συμβουλίου, η Δανία έκανε ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει αυτές τις πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερα στο θέμα λοιπόν του, των πρωτοβουλειών που ανέλαβε η Δανία στο Κάτεγκατ. Ε, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο να αναλαμβάνει πρωτοβουλίε, να ενημερώνει τα υπόλοιπα κρατημέλη για τέτοιου τύπου ε, εξελίξει. Πώ είναι δυνατόν τέτοιε συζητήσει να γίνονται με μυστικότητα. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και θα πρότεινα στην Επιτροπή να συνεργαστεί με εμά έτσι ώστε αυτά τα πράγματα να έρχονται στο φω τη δημοσιότητα. Όπω για παράδειγμα αυτά που. Τι λανθασμένε επιλογέ που έκανε η Δανέζικη κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσουμε το λόγο στα άλλα μέλη της Επιτροπής, ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή της ΕΟΚΕ, τον κύριο Σίμονς, ε, για να συνεισφέρει στη συζήτηση. Έχετε τρία λεπτά. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Συμφώνησα με την γραμματεία δύο λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Με χαρά άκουσα αυτά που πρότειναν ε, οι βουλευτές για την έκθεση και γι' αυτό λοιπόν θα είμαι σύντομος. Ότι συμφωνούμε με πολλά από τα στοιχεία που σε έχει συμπεριλάβει ο εισηγητή στην έκθεση. Την ίδια κατεύθυνση ακολουθούμε και εμεί ε, προσυπογράφουμε λοιπόν από την Επιτροπή μας ε, τα θέματα αυτά και έχουμε ε, προσωπογράψει μάλλον ένα ε, κοινό έγγραφο σε ό,τι αφορά τους ωκεανούς, παρά το γεγονός ότι ασφαλώς έχουμε κάποιες παρατηρήσεις να κάνουμε. Μία εκ των πιο σημαντικών είναι ότι και εδώ θα πρέπει να αντιληφθούμε τον κατεπίγοντα χαρακτήρα ο εισηγητής ε, προφανώς αναφέρει και την επιβολή σαφώνα ε, προθεσμιών. Και από πλευρά τη Επιτροπή ε, σκοπεύουμε να εργαστούμε τάχιστα για το θέμα αυτό. Να αξιοποιήσω το υπόλοιπο χρόνο που έχω στην διάθεσή μου για να τονίσω τα τρία σημεία τα οποία δεν τα βρήκα να αποτυπώνονται στην έκθεση. Να αναφέρω κάποια σημεία από την γνωμοδότηση προκειμένου να είναι πιο απλό και για τον σκιωδή και για τους κοιόδες και για τον γιατί να τα παρακολουθήσουν. Αφορά το σχετικό Ευρωπαϊκό Φόρουμ, γιατί πρόκειται για ένα οριζόντιο θέμα και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να έχουν ε, επιρροή εδώ για να δούμε το πότε, πώς και με ποιον τρόπο θα πετύχουν αυτά Ύστερα, σε ό,τι αφορά το μυθμένο της θάλασσας, προτείνουμε να υπάρχουν στοχευμένες αξιολογήσεις, όπως γίνεται και επί ξηράς, σε ό,τι αφορά τις σχετικές αξιολογήσεις, γιατί να μην γίνει το ίδιο και με το μυθμένα της θάλασσας. Και τέλος, κάτι που επίσης αναφέρεται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μάλλον ούτε στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε στο δικό σας έγγραφο, για ευκαιρίες απασχόλησης. Θα ήταν ε, πραγματικά ωφέλιμο να μπορούσε να βρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα σήμαινε αυτό για θέματα εκπαίδευσης προσόντων και να κλείσω επαναλαμβάνοντας ότι αυτά τα στοιχεία μας απασχολούν και θα θέλαμε να τους δοθεί ιδέουσα προσοχή. Ευχαριστούμε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ και γιατί τηρήσατε το χρονοδιάγραμμα με τόση ακρίβεια. Και τώρα να περάσουμε στα μέλη της Επιτροπής ε, για να ακούσουμε τα σχόλιά τους. Πρώτα η κυρία Ντάλη, σας παρακαλώ δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ε, ευχαριστώ στον εισηγητή για τις αρχικές καλές παρατηρήσεις τις οποίες μας παρουσίασε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε τρεις τομείς οι οποίοι κατά την άποψή μου ε, μαζί άλλωστε με το σκιώδη συγητή των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, θεωρούμε ότι πρέπει να φροντίσουμε περισσότερο, κυρίως τις εκπομπές και τις εκπομπές των σκαφών και εδώ θα συμφωνήσω με την άποψη του σκιώδη συγητή μα ότι πρέπει ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τονίσουμε την ανάγκη να παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια στους, στα σκάφη, στου Ευρωπαϊκού λιμένε, αυτή τη στιγμή μπαίνουν στο λιμάνι. Έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε τη ρήπανση στους λιμένες μα, διότι τα σκάφη θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν τι ε, μηχανές του ε, και θα χρησιμοποιούν ε, ενέργεια η οποία θα παρέχεται από τους λιμένες θα υποβάλω και σχετικές τροπολογίες ώστε να ε, τονίσουμε και τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG στα σκάφη, που είναι πολύ πιο ε, καθαρό κατά την άποψή μου από αυτό που σημαίνει, συμβαίνει αυτή τη στιγμή και τα επίπεδα ρήπανσης που δημιουργούν τα σκάφη, κυρίως ε, στις θάλασσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι το θέμα των θαλασσίων απορριμμάτων, διότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί που μας περιβάλλουν σύντομα θα περιλαμβάνουν ένα τόνο απορριμμάτων για κάθε τρεις τόνους ε, ηχθείων και αυτό θα συμβεί σε λιγότερο από 10 χρόνια από σήμερα. Θα υποβάλουμε λοιπόν και κάποιες προτάσεις ε, για πρωτοβουλίες ώστε να αντιμετωπιστεί το σχετικό ζήτημα. Και κάτι τελευταίο. η ανάγκη να σταθούμε περισσότερο στον τομέα της έρευνας, διότι ο μετριασμός των συνεπειών του κλίματος ε, βασίζεται και σε αυτές τις πολιτικές. Εμείς λοιπόν ως Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα θέματα αυτά, διότι μπορούμε να τα τονίσουμε περισσότερο και έχουμε δυνατότητες ε, να ε, υποστηρίξουμε τις πολιτικές μας για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, ιδίως όσον αφορά το κλίμα για τις δράσεις αυτές. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει το συντομότερο δυνατόν τις δυνατότητες του Κοπέρνικους για τη μέτρηση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου, κυρίως του διοξιδίου του άνθρακα, διότι αυτό θα έχει μεγάλη αξία και θα έχει και αντίκτυπο στην μάχη που δίνουμε για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Ο κύριος Φλόρεντς τώρα για δύο λεπτά αυτό. Äh, Σα ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον εισηγητή και πραγματικά υποστηρίζω το όσο μας είπατε. Αλλά θα ήθελα να βάλουμε λίγο ξύδι στο κρασί μας. Γιατί κάνουμε λες και μόλις ξεκινήσαμε με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μα 20 χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και καταγγέλλεται και δικαίω ότι τα λύματα κατά 80% είναι από τη ξηρά. Αναρωτιέμαι πού βρίσκονται τελικά, ποια κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία δεν εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προκειμένου να μην καταλήγει αυτό το 80% στι θάλασσε. Τώρα να κάτσουμε να γράψουμε ένα καινούριο έγγραφο και να, τα, να θεωρήσουμε ότι έτσι το έχουμε ρυθμίσει το θέμα, είναι πραγματικά απλάνη. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αν δεν έχουμε το θάρρο και την τόλμη, επιτέλου να εφαρμόσουμε στην Ευρώπη και στις, ε, στα κράτη-μέλη τα όσα έχουμε αποφασίσει πριν από πολλά χρόνια. Δεν καταλαβαίνω πώς πιστεύετε ότι με ένα καινούργιο αριθμητικό στοιχείο θα αλλάξει οποιαδήποτε κατάσταση, θα υπάρξει οποιαδήποτε κίνηση. Μα η νοοτροπία στο κεφάλι μας πρέπει να αλλάξει πρώτα. Δεν έχω καμία όρεξη μετά από 28 χρόνια να ψηφίσω τον ιωστό έγγραφο και τελικά να μην αλλάξει τοτεδήποτε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, ε, είσαστε νέος και δεν έχετε ακόμα κουραστεί αλλά να σας πω ότι έχω καλήσει τις πρεσβείες που δεν τηρούν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αλλά τελικά καταλήξαμε σε μια τεράστια διαμάχη. Μα ακριβώς αυτή τη μάχη πρέπει να δώσουμε. Να τσακωθούμε πρέπει. Και με την κυρία, τη συνάδελφο από την Δανία, όπως τη λένε την κυρία Άουκεν. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να αντισταθούμε, να παλέψουμε. Είμαστε πολύ ε, καλοί μαθητέ. Ε, κάνουμε τα μαθήματά μας, γράφουμε ένα καινούργιο έγγραφο και θεωρούμε ότι θα αλλάξει το οτιδήποτε. Μα τίποτα δεν θα αλλάξει, τίποτα δεν θα έχει ρυθμιστεί. Ευχαριστώ. Μακάρι να ήμουν και εγώ τόσο νέο όσο πιστεύετε, αλλά τέλο πάντων να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Κυρία ευχαριστώ. πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να προσέξουμε το θέμα των ωκεανών, αλλά άκουσα και μερικά ζητήματα να φύγονται που θα ήθελα να ανασχολιαστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την ε, μόλυνση από τα λοιπάσματα, από τη γεωργία. Από πού συλλέγουμε τα στοιχεία αυτά, τα αριθμητικά στοιχεία αυτά, γιατί άκουσα, για παράδειγμα, από την Επιτροπή μας ότι ε, μειώθηκαν ε, τα τα φωσφορικά άλατα και τελικά δεν υπάρχει ε, ε απαρκής ποσότητα φωσφορικών αλάτων. Και κατά δεύτερον, ε, επιλεκτική και βιώσιμη αλία σε ό,τι αφορά τον τρόπο που γίνεται η αλία και κυρίως πώς διαμορφώνεται η βιώσιμη αλία και πώς αυτό επηρεάζει τους ωκεανούς. Και ελπίζω ιδιαίτερως, επιτρέψτε μου να πω ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη διαδικασία αυτή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Κοινοβουλίο, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλο όγκο πρωτοβουλειών που αξίζουν τι υποστηρίξει μα. Ευχαριστώ πολύ. Και δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο. Επομένω, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Παπακουσταντίνου έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Φαρία, για το σχέδιο εκθεσής του και τα μέλη της Επιτροπής για τα επικοδηματικά του σχόλια. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ύπατη εκπρόσωπος ε, δημοσιεύουν μια δήλωση πολιτικής ε, αυτής της μορφής για τους ωκεανούς. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ μεγάλο άλμα και επειδή ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές το επεσήμαναν, ε, το διεθνές πλαίσιο παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολύ καλή ευκαιρία να εξασφαλίσει ότι θα πρωτοστατήσει σε πολλά θέματα, όπως για παράδειγμα την κλιματική αλλαγή και τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Η το Διεθνές Θεματολόγιο για τους ωκεανούς είναι τμήμα των δεσμεύσεών μας για το 2030, κυρίως ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης 14. Θα ήθελα να σας παραπέμψω στην πρόσφατη ε, διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία έγινε ε, νωρίτερα εντός του μηνός ε, και είχαμε συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Φαρία ήταν επικεφαλής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συγκεκριμένη διάσκεψη ε, αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην δημόσια συζήτηση σε διεθνές επίπεδο για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τους ωκεανούς μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ε, πολύ μεγάλες δεσμεύσεις ε, στη συγκεκριμένη διάσκεψη και ο στόχο μα είναι να διατηρήσουμε αυτή την ουσιαστική ορμή που δημιουργήθηκε και φέτος ε, στη Μάλτα στις 5 και 6 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φιλοξενήσει μια μεγάλη διεθνή διάσκεψη για τους ωκεανούς. Με αυτή την ε, διεθνή ανακοίνωση για τη διακυβέρνηση των ωκεανών ε, καθορίζουμε ένα συγκεκριμένο θεματολόγιο που θα βασίζεται σε δράσεις σε τρεις ε, τομείς προτεραιότητες. Πρώτον, να βελτιώσουμε το πλαίσιο διεθνούς διακυβέρνηση των ωκεανών. Έτσι θα αναβαθμίσουμε τις προσπάθειές μας για την έγκριση, κύρωση και αποτελεσματική εφαρμογή βασικών μέσων για τη διακυβέρνηση των ωκεανών και θα εξετάσουμε με βιώσιμο τρόπο πώς μπορούμε να προωθήσουμε και να ε, υλοποιηθεί το σχέδιο ε, της Άγκλος ε, για τη διεθνή δικαιοδοσία. Ε, όσον αφορά τη δεύτερη προτεραιότητα, να μειώσουμε τις ανθρώπινες πιέσεις στους ωκεανούς, ε, θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις πιέσεις στους ωκεανούς, όπως για παράδειγμα ε, ρήπανση των θαλασσών λόγω της κλιματικής αλλαγής και να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ωκεανοί και η βιοπικιλότητά τους. Και ο τρίτος τομέας προτεραιότητας που είναι η ενίσχυση των διεθνών δεδομένων και της συνεργασίας θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τις γνώσεις μας για τους ωκεανούς. Οι θαλάσσιες τεχνικές ε, μας προσφέρουν νέες δυνατότητες και θέλουμε να τις εκμεταλλευτούμε. Όσον αφορά την ερώτηση ε, της κυρίας Άουκεν, θα ήθελα να πω ότι η στρατηγική για τα πλαστικά θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλη του έτους και στην στρατηγική για τα πλαστικά θα ε, προσθέσουμε και την αναθεώρηση της ε, οδηγίας ε, για τη διαχείριση των αποβλήτων. Και όσον αφορά την εξόριξη ε, στον βυθό της θάλασσας. Αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, προσελκύει όμως ιδιαίτερα ενδιαφέρον διεθνώς. Ο ISA ολοκληρώνει τον κώδικα εξόριξης ε, για την εκμετάλλευση των πόρων. Παρακολουθούμε στενά τα όσα διαδραματίζονται στο συγκεκριμένο βήμα και υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας και θα συζητηθούν εκεί. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει σε μια σειρά από προγράμματα μαζί με τα κράτη-μέλη και ε, τον πανεπιστημιακό τομέα, ερευνητικά Ινστιτούτα και Ιδρύματα επίσης ε, για αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα και ένα από τα βασικά προγράμματα είναι το πρόγραμμα Μίδας. Ε, ένα ουσιαστικό στοιχείο για μας στο θέμα αυτό είναι ότι όλες οι δράσεις που σχετίζονται με ωκεανούς, είτε πρόκειται για τα απορρίμματα, για την κλιματική αλλαγή, για τους πόρους κλπ, αποτελούν ε, τμήμα μιας ολιστικής προσέγγισης. Οι πιέσεις που υπόκειται οι ωκεανοί είναι αλληλένδετες και οι λύσεις που πρέπει να παρέχουμε θα πρέπει να είναι και αυτές αλληλένδετες. Η επιτυχία της δράσης μας εξαρτάται και από τη δέσμευσή μας με διεθνείς εταίρους, διότι πρόκειται για παγκόσμια πρόκληση και μία από τις βασικές δράσεις ε, που προωθεί η ανακοίνωση είναι να υπάρχουν εταιρικές συμπράξεις ε, για τους ωκεανούς ε, με χώρες κομβικές και αυτό αναφέρθηκε και από τον εισηγητή και από τους κοιόδης εισηγητές και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, με την ανακοίνωση αυτή ε, παρουσιάσαμε τη φιλοδοξία μας να διαδραματίσουμε κεντρικό ρόλο στην σωστή διαχείριση των ωκεανών. Έχουμε ήδη λάβει υποστήριξη από το Συμβούλιο που ενέκρινε τα συμπεράσματά του για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών τον Απρίλιο. Το Συμβούλιο απέστειλε ένα πολύ θετικό μήνυμα για να προχωρήσουμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως βασικό εταίρο σε αυτή την ε, τεράστια προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσω και πάλι το λόγο στον εισηγητή για να ε, συνοψίσει. Έχετε το λόγο κύριε Φαρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις σας. Ε, σημείωσα ε, ό,τι άκουσα. Προφανώς και υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανησυχίες, ε, τις οποίες ακούσαμε και εδώ. Θα ήθελα να συμπεριληφθούν και στο κείμενο Βεβαίως πολλά από αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο κείμενο ήταν καρπός ε, διαπραγμάτευσης μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα βέβαια να είχαμε πάει έτσι περαιτέρω. Ε, έλαβα ε, στοιχεία από τους συναδέλφους, ε, συνεχίζω να λαμβάνω τη συμβολή τους και ελπίζω να μου δώσουν και στη συνέχεια στοιχεία, διότι το κείμενο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Σίγουρα θέλουμε να έχουμε κάτι λογικό, το οποίο όμως ακόμα πρέπει να διευκρινιστεί. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, όπως αυτά που αναφέρθηκαν εδώ σήμερα. Σημείωσα πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα αναφερθώ βέβαια εδώ σε όλα τα στοιχεία. Υπάρχει ένα νέο όρομα, όπως ακούστηκε, θα ήθελα να σας πω ότι ένα από τα θέματα που με απασχολεί ιδιαίτερως είναι ε, το θέμα των εκπομπών των ε, θαλασσιών μεταφορών και όλες οι εκπομπές, όχι μόνο οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Όπως ξέρετε, ήμουν εισηγητής και σε μια άλλη έκθεση για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για τις θαλάσσιες μεταφορές και εκεί θα ήθελα να είχα πάει πιο πέρα, αλλά δεν τα κατάφερα. Ελπίζω να μπορέσουμε να αυξήσουμε το επίπεδο με το έγγραφο αυτό και να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει στο μέλλον. Στι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα θα είμαι στην, ε, στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στο Λονδίνο και ένα από τα θέματα ε, τα οποία θα θίξω θα είναι αυτό. Επίση, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλου, Όπως σας είπα, σημείωσα πάρα πολλά πράγματα, αρκούν αυτά για να κάνω αλλαγές, ε, τις οποίες θα παρουσιάσω σε όλους. Αυτά λοιπόν, ευχαριστώ τους συναδέλφου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φαρία. Και τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 5 Ιουλίου, 11 η ώρα. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Τραν στις 25 Σεπτεμβρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΜΒΗ 28 Σεπτεμβρίου. Και στην Ολομέλεια θα ψηφιστεί στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Ακόμα είναι προσωρινή βέβαια αυτή η ημερομηνία. Περιμένουμε όμως ε, ότι θα υπάρξει ψηφοφορία στη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και περνάμε στις ψηφοφορίες. Έχουμε μια ψηφοφορία για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ε, Κινητικότητα Χαμηλών Εκπομπών. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Τζόφολη. Αν είστε έτοιμοι και έχετε τις κάρτες σας και λειτουργούν και όλες. Ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση. Επαλήθευση λοιπόν για τη συμβαστική τροπολογία 17. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 75. Ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 80 και 270 είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αμποχές, νομίζω απορρίπτεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. Πέρας Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 δεν ψηφίζουμε, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ΤΡΑΝ. Πάμε στην 96 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 109 όχι, καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112 υπέρ. Σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ. Κατά, αποχές, επαλήθευση. Vote is closed. Adopted. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Α ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Παρακαλώ. Πέρα ψηφοφορία εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές το ίδιο με πριν εγκρίνεται λοιπόν συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 137 και 142 είναι ίδιες, παρακαλώ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 138 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο 141 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16. Υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε την 144. Μάλιστα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 168 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 169 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 170 υπέρ, κατά αποχές θα την ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ για την 170. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μου φάνηκε ότι υπορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 200. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 208. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 216 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 218 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 246 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 22. Να ελέγξουμε θέλετε για την 246. Ψηφίστε παρακαλώ. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 271 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 272 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 273 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Υπέρ της ψηφορίας. Εγκρίνεται. 275 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 277 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε καλύτερα ψηφίστε παρακαλώ εγκρίνεται με μικρή διαφορά Όχι, δεν αλλάζει κάτι. 278 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 279 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 280 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε. Εγκρίνεται 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 36 υπέρ. Κατά. Α, όχι, να ελέγξουμε την 35 θέλετε. Ναι. Ψηφίστε παρακαλώ για την 35. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με την ίδια πλειοψηφία όπως και πριν. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά, η κλίση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Thank Όσοι επιθυμείτε να φύγετε μετά την ψηφοφορία, παρακαλώ να φύγετε τώρα, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Σημείο νέα. Έκθεση Γκροστέτ για το έλεγχο αναλογικότητα πριν από την, νέα έγκριση, από την έγκριση του νέου κανονισμού για τα επαγγέλματα. 30 δεύτερα σας δίνω, όσοι επιθυμείτε. Όχι 30 λεπτά, 30 δευτερόλεπτα. Προτιμάτε 30 λεπτά. Good. Okay. It's Dali. Dali. Yeah. Good. Then we continue our... Πολύ ωραία, να συνεχίσουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Να επικεντρωθούμε στο επόμενο σημείο, το οποίο είναι η έκθεση Γκροστέτ και θα ήθελα να δώσω κατευθείαν ε, τον λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Γκροστέτ. Γιατί το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε λοιπόν μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θέλει να υλοποιήσει μια διαθρωμένη διαδικασία για έναν έλεγχο αναλογικότητα σε ό,τι αφορά τα νέα μέτρα τα οποία εγκρίνονται από τα κράτη-μέλη ε, για να ρυθμίζονται τα διάφορα επαγγέλματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ε, την οτροπία και το σκόπο που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συναντηθήκαμε και με εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι ο ειδικό χαρακτήρα των επαγγελμάτων στον τομέα τη υγεία σε ό,τι αφορά το δημόσιο λειτουργήμα το οποίο επιτελούν και εδώ υπογραμμίζουμε ε, στο θέμα αυτό, δεν λαμβάνεται παρκώς υπόψη στο σχέδιο της ε, οδηγία και ως εκ τούτου προτείνω να εξαιρεθούν αυτοί οι τομεί από το πεδίο εφαρμογή. Σήμερα τα κράτη-μέλη ήδη στο πλαίσιο του άρθρου 59 της οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν για την προστασία κάποιων επαγγελμάτων τα οποία είναι αναλογικά. Και μιλάμε πάντα για τέτοια επαγγέλματα για τα οποία χρειάζεται άδεια, τα προστατευμένα. Και λοιπόν, ε, ο τομέας της υγείας υπάγεται στην άσκηση αυτή, στο πεδίο εφαρμογή του άρθρου 59 της ε, οδηγία για τα συγκεκριμένα προσόντα. Ωστόσο, θεωρώ ότι θα περάσουμε σε μία εξπόστα ε, αξιολόγηση και θα πρέπει να περνάμε να περάσουμε από μία εξπόστα σε μία εξάντε τέτοια δικασία αξιολόγησης, γιατί είναι πολύ γραφειοκρατική και περίπλοκη διαδικασία. Αυτό συχνά το κατηγορούμε, το επιρρύπτουμε ως ευθύνη κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, προφανώς ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξηγεί ότι δεν έκανε παρακωδικοποίηση των εφιστάμενων κανόνων προκειμένου να ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις για όλους και να μην υπάρχουν νομικές διαφορές και προσαγωγές στο δικαστήριο. Καταλαβαίνω φυσικά το σκοπό αυτό. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκεί που διαπιστώνει ότι υπάρχει νομική αβεβαιότητα, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας θεωρούν ότι υπάρχει ευελεξία για τα κράτη-μέλη. Έτσι ερμηνεύουν αυτή την αβεβαιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτό επιτρέπει στα κρατη να προσαρμόσουν στις τοπικές ιδιότητες τον κλάδο αυτό. Και παρεπιπτόντω, ε, αυτό έχει αποφαθεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην ομολογία του. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί σα ε, ε, ομολογώ ότι κατανοώ ποιε είναι οι προθέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά κοιτάξτε, δεν μα λείπουν οι καλέ προθέσει. Αλλά όλα αυτά μπορεί να πετύχουμε ε, κακά αποτελέσματα. Και σε ό,τι αφορά το άρθρο 59 της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα, μου φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά καταλήγει να υλοποιεί μια διαδικασία πάρα πολύ περίπλοκη με ένα σωρό εξαιρέσεις για τον τομέα της υγείας, αλλά τελικά δημιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ περιοριστικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν με την πρόταση αυτή ουσιαστικά αποτρέπει τα κράτη-μέλη να υλοποιούν προδιαγραφές για τον τομέα της υγείας προσαρμοσμένες στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοί σας προτείνω να προσαρμοστείτε το πεδίο εφαρμογής και να εξαιρεθούν τα επαγγέλματα στον κλάδο της υγείας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει και πρόεδρος και τώρα να δώσουμε το λόγο στους κοιόδες εισηγητές. Να σας ζητήσω να μην ξεπεράσετε τα τέσσερα λεπτά ως σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία Ντάλη είναι η πρώτη από τους σοσιαλδημοκράτες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και να σας πω ότι α, αντικαθιστώ την κυρία Τζεντήλα η οποία είναι η σκιώδης εισηγήτρια για το θέμα αυτό και τη δική σας θέση θα παρουσιάσω σε ό,τι αφορά την γνωματοδότηση αυτή. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για το σχέδιο γνωματότησης και σημειώνουμε ασφαλώς την τοποθέτηση της εισηγήτριας, να εξαιρεθούν δηλαδή όλα τα επαγγέλματα του τομέα της υγείας, δεδομένου της φύσης ε, του λειτουργήματος και παράλληλα όμως ως ομάδα εξετάζουμε τη λύση αυτή και γίνονται και σχετικές συζητήσεις στην ομάδα μας και θα συνεχίσουμε από αυτές τις θέσεις ε, στην ομάδα μας στη συζήτηση. Η ίδια η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα θέτει την αρχή και τις προδιαγραφές αναλογικότητας και εδώ συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας. Άρα αυτό που προτείνει η συγγητρία είναι μια εξαίρεση της εξαίρεσης και κατανοώ ότι οι σχετικές ευρωπαϊκές οργανώσεις που καλύπτουν και τους οβοντιάτρους και τα υπόλοιπα ιατρικά επαγγέλματα ανησυχούν σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης όπως περιλαμβάνεται στην οδηγία και επικαλούνται ε, λόγους δημόσιας υγείας, προστασίας των ασθενών και κατανοούμε ότι αυτό τώρα ήταν θέμα των κρατών μελών και τα κράτη-μέλη αυτή η οδηγία θα έχει επιπτώσεις και θα επηρεάσει και την αρχή της επικουρικότητας στο πλαίσιο αυτό. Ωστόσο, θα θέλαμε να εκφράσουμε και την τοποθέτηση της έκθεση ΣΒΑΜΠ, η οποία συντόμως θα δημοσιευθεί και ως ομάδα θέλουμε να τοποθετηθούμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τελικά αυτή η οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας τελικά θα πετύχει τα όσα επιδιώκουμε. Και θα καταθέσουμε και τροπολογίες εν χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής από την ομάδα της Άλτε, η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ αντικαθιστώ την κυρία Μούλερ, που είναι η σκιώδη εισηγητρία, η οποία δυστυχώ δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν, εξ ονόματος τη κυρία ε, Μουλερ, την κυρία Κροστέτ και να πούμε ότι υπάρχουν και κάποια ζητήματα τα οποία όντω ε, τα θέματα μάλλον τα οποία επικαλείται η συγγήτρια είναι προφανώ τα πιο βασικά στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ό,τι αφορά του περιορισμού. Ε, σε κάποια επαγγέλματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά για να εξασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Η οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσφόντων ζητά να υπάρχει έλεγχο αναλογικότητα για τα μέτρα αυτά, γιατί η εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει κάποιες, ε, κάποια ελλείμματα. Η πρόταση λοιπόν ε, θέλουμε να καταλήξει σε μια οδηγία για πιο πολύ σαφήνεια και καλύτερη υλοποίηση. Από πλευρά τη Επιτροπή μα όμω πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιε βελτιώσει σε κάποια σημεία. Καταρχά, τα επαγγέλματα στην τομέα της υγείας δεν είναι κλασικά επαγγέλματα. Οι ασθενείς δεν είναι καταναλωτές με την παραδοσιακή έννοια. Θα πρέπει να γνωρίσουμε αυτόν τον ιδιαίτερο ρόλο των επαγγελμάτων αυτών. Και η Ρίκ Μούλερ λέει κάτι διαφορετικό ότι, από αυτό που πιστεύω εγώ στο θέμα αυτό για το κατά πόσο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογή. Και τώρα θα συνεχίσουμε με την τοποθέτηση τη Ούλη και Μιούλερ. Κατά δεύτερον, η οδηγία θα πρέπει να οδηγήσει σε καλύτερη υλοποίηση του, ελέγχου αναλογικότητα. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι όταν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση για λόγου προστασία του καταναλωτή και δημοσία υγεία, δεν μπορούν να επιβαρυνθούμε επιπλέον γραφειοκρατία. Εκτό αυτού, δεν μπορούν να επιβαρυνθούν και αυτοί οι οποίοι ήδη εφαρμόζουν σωστά την αρχή της ε, λογοδοσίας. Και ακόμα και αυτός ο έλεγχος αναλογικότητας θα πρέπει να είναι αυτού αναλογικός. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εκ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφη, Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο που μας παρουσίασε σε ό,τι αφορά τις αμφιβολίες για τον τομέα των επαγγελμάτων στον τομέα της υγείας θα πρέπει να εμβαθύνουμε από πλευρά τη ομάδα μα. Εγώ έχω να σα πω το εξή: 22% των Ευρωπαίων εργαζομένων ε, εργαζόνται σε κατοχυρημένα επαγγέλματα. 15 εκατομμύρια άνθρωποι λοιπόν από τον αριθμό και μόνο κατανοούμε πόσο μεγάλη είναι η έκταση και ποιες είναι οι συνέπειες της έκτασης αυτής η ευρωπαϊκή εφαρμογή της εξάντε αξιολόγησης αναλογικότητας ε, θα ωφελούσε ιδιαίτερα τους νέους που θέλουν να κινηθούν προς το εξωτερικό και τις ευρωπαϊκές ιδέες. Θεωρώ ότι με την έκθεση αυτή υποστηρίζουμε και ενισχύουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι προστατεύουμε και από περιβολικό προστατευτισμό τα επαγγέλματα αυτά. Τα ρυθμιστικά εμπόδια τα οποία περιορίζουν την έναρξη σε τέτοια επαγγέλματα θεωρώ ότι θα οδηγούσαν τις τιμές ε, στα ύψη. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι να ταχθούμε υπέρ της ελεύθερης μετακίνησης των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια βασική προϋπόθεση είναι η δυνατότητα οι εργαζόμενοι σε όλα τα κράτη-μέλη να μπορούν να ασκούν το επάγγελμα στο οποίο έχουν καταρτιστεί. Και αυτό να με τον πιο απλό δυνατό τρόπο. Πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά τις εθνικές προδιαγραφές είναι προτιμητέα η κατάσταση αυτή σε σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Αϊκάουτ. Uh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης και τις τρεις τροπολογίες. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη συζήτηση που θα κάνουμε είναι κατά πόσον θα αποκλείσουμε ή όχι τα ιατρικά επαγγέλματα. Εμείς ως πράσινοι, για να είμαστε ειλικρινείς, είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βλέπουμε τώρα ότι η συγγήτρια προτείνει μια εξαίρεση, την οποία εξετάζουμε. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, ίσως θα μπορούσε λοιπόν η συγγήτρια να μας πει λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε και εμείς τη θέση μας. Ε, σαφώς, ε, όπως είπε και η κυρία Ντάλη, υπάρχει σχέση μεταξύ της οδηγίας ε, ε, αυτής και της οδηγίας για τα επαγγελματικά ε, προσόντα, στην οποία δεν αποκλείονται τα ιατρικά επαγγέλματα. Έχουμε λοιπόν δύο οδηγίες, στην οποία στη μία θα αποκλείονται και στην άλλη όχι. Μήπως είναι κακή νομοθέτηση αυτή. Δεύτερον, δεν είμαι βέβαιη ως τι ακριβώς προσπαθεί να επιτύχει η συγγήτρια με αυτή την εξαίρεση τι ακριβώς ε, πιστεύετε ότι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη τώρα, τα οποία δεν θα μπορούν να γίνουν ή θα είναι πολύ πιο δύσκολο να υλοποιηθούν μέσω αυτής της οδηγίας. Επίσης, υπάρχει ένα άρθρο 5 εδώ, βάσει του οποίου τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν στόχους δημοσίου συμφέροντος για να αλλάξουν ε, τη ρύθμιση κάποιων επαγγελμάτων. Επομένως, το άρθρο 5 ούτως ή άλλως δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να το χρησιμοποιήσουν αυτό. Γιατί λοιπόν να αποκλείσουμε έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο. Αυτά τα ερωτηματικά μας δημιουργούνται. Προσβλέπουμε λοιπόν τις απαντήσεις της εισηγήτριας. Τι πιστεύετε λοιπόν ότι θα μπορούσε να ε, μην επιτρέπεται ουσιαστικά στα κράτη-μέλη από την οδηγία και γιατί να ε, επιλέξουμε αυτή την εξαίρεση. Και τώρα όσον αφορά κάποια τελευταία στοιχεία. Εμεί είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υποβάλουμε τροπολογίε μόνο για το άρθρο 7 για τη διαβούλευση των εμπειρογνωμόνων και τη διαφάνεια στο άρθρο 9 για να τα βελτιώσουμε αυτά, αλλά θα είναι ίσονα σημασία. Κατά τα λοιπά, είμαστε ικανοποιημένοι με την οδηγία όπω προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσβλέπουμε φυσικά και στη συζήτηση με του κοιόδη συγητέ και ε, με την εισηγήτρια, κυρίω ε, για το κατά πόσον θα δεχτούμε ή όχι την εξαίρεση για τα ιατρικά επαγγέλματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχουμε τα μέλη της Επιτροπής. Τρία λεπτά ο καθής. Ο κύριος Λίζε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω ιδιαίτερα στην πρόταση της Φρανσουάς Γκροστέτ και πιστεύω ότι επικρατεί μεγάλη ανησυχία στα ιατρικά και παραγιατρικά αυτά επαγγέλματα σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη επιβολή παραπάνω γραφειοκρατία και νομίζω ότι η Φρανσουάζ έχει ήδη απαντήσει την ερώτηση του κυρίου Άικχατ. Θα κάνουμε μια εκ των προτέρων ε, αξιολόγηση αν αποδεχτούμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο έχει και δεν πιστεύουμε ότι αυτό θα πετύχει επαρκή αποτελέσματα για να δικαιολογήσει όλη την αναστάτωση που θα προκαλέσει. Δεν υπάρχει κάποιο πιστικό λόγο ε, για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώ και ο Ανδρέας Σφαμπ, ο εισηγητής στην ε, καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, κάτι παρόμοιο προτείνει και νομίζω ότι θα πρέπει να το ακολουθήσουμε ως πρόταση. Αν μας αποδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι ανησυχίε μας δεν είναι βάσιμες, το ξανασυζητάμε. Αλλά μέχρι τότε πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ σόφρονες σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό και να ακολουθήσουμε την πρόταση της Φρανσουάς ε, Γκρουστέτ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπως την υπέβαλε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. κύριε Ντόρφμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι επί της αρχής θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα θέματα του, τα επαγγέλματα του υγειονομικού κλάδου είναι επαγγέλματα όπου υπάρχουν ε, εμπόδια σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή εργατικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτά θα πρέπει να καταληθούν. Και αυτό μόνο εν μέρη δικαιολογείται θεωρώ ότι υπάρχουν αυτά τα εμπόδια. Μιλάμε για κατάρτιση, για νοσοκομιακό προσωπικό, για του γιατρού. Θα σα πω τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την πρόταση αυτή, αλλά ένα Ιταλό γιατρό στη Γερμανία ε, ακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτιση, επέστρεψε στην Ιταλία και τώρα του δεν το αναγνωρίζονται οι τελικοί εξετάσεις στη Γερμανία, γιατί δεν βρίσκεται στη Γερμανία πλέον και δεν είναι εγγεγραμμένο ε, στα γερμανικά μητρώα. Είναι πραγματικά παράλογο και νομίζω ότι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα επαγγέλματα του υγειονομικού κλάδου θα πρέπει να κοιτάξουμε το τι είναι δικαιολογημένο και τι δεν είναι δικαιολογημένο, τι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ασθενή και τι όχι. Τι αποτελεί απλά εθνική, εθνικό περιορισμό που πολύ απλά έχει ως σκοπό να προστατεύσει την εθνική αγορά και νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και τη δεύτερη κατηγορία αυτή και να βρούμε και λύσεις σε ό,τι αφορά και το γεγονός ότι ακριβώς τα επαγγελματα αυτά του υγειονομικού κλάδου έχουν μεγάλη ζήτηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό λοιπόν έχει νόημα η ανταλλαγή εργατικού δυναμικού στα επαγγελματά αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάντεμπαχ. Ευχαριστώ. Και εγώ, όπως είπε η κυρία Αγροστάτ, πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για, τον, ε, για την εξαίρεση των επαγγελματών αυτών από τα πεντή εφαρμογή. Όπω είπε και η κυρία Ντάλη, θα το συζητήσουμε αυτό επισταμένω και στην πολιτική μα ομάδα. Γιατί στην παρούσα φάση φαίνεται ότι θα ήταν πλεονέκτημα να εξαιρεθούν από τα πεντή εφαρμογή τα επαγγέλματα αυτά. Θα ήταν προ το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Σε ό,τι αφορά δηλαδή την, τον έλεγχο αναλογικότητα. Και νομίζω ότι σίγουρα θα πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό τι επόμενε εβδομάδε στην ομάδα μα. Ευχαριστούμε. Και τώρα να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλα τα κράτη-μέλη για τις απόψεις που εξέφρασαν. Δεν θα σας εκπλήξει βεβαίως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ικανοποιημένη για την υποστήριξη και την αναγνώριση από αρκετά μέλη ότι οι υπηρεσίε της υγείας σίγουρα θα έχουν θέση σε αυτή την πρόταση. Ο κύριος Λίζε ζήτησε και κάποια ε, εξασφάλιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μπορώ να σας δώσω όσες εξασφαλίσεις θέλετε και πολύ ευχαριστώ να σας δώσω και άλλες αν θέλετε να προχωρήσουμε. Πρώτον, καταρχάς τα ιατρικά επαγγέλματα είναι σημαντικό τμήμα της οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα. Αναθεωρήθηκε το 2013 σχετική οδηγία και ο νομοθέτης, εσείς δηλαδή και οι συνάδελφοί σα. Και ο στόχος είναι να είναι αναλογική η οδηγία, δηλαδή επιτελεί το σκοπό για τον οποίο ε, ε, συστάθηκε, κυρίως προστασία της υγείας βεβαίω, αλλά δεν υπερβαίνει τα όσα είναι απαραίτητα για την επίτευξη αυτή του στόχου και δεν δημιουργεί περιτά προσκόμματα για ελεύθερη κυκλοφορία, για νέους ε, πτυχιούχους και για πρόσβαση στο επαγγελμά. Και επίσης και για τους ίδιους επαγγελματίες για την άσκηση του επαγγελματός τους. Αυτή η διαδικασία ε, που εισάγεται από την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα καθορίστηκε με τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη εξέτασαν όλη την κείμενη νομοθεσία, θα έλεγα σχεδόν όλη την κείμενη νομοθεσία. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη σε κάποια επαγγέλματα στα οποία δεν έχουμε λάβει ακόμα τι απαραίτητε πληροφορίε και την αξιολόγηση περί αναλογικότητα. Αυτά για την κείμενη νομοθεσία, τα οποία περιλαμβάνουν βεβαίω και τα ιατρικά επαγγέλματα. Ε, τώρα, Βάσει των πληροφοριών που είδαμε και λαμβάνοντα υπόψη και τι κατευθυντήριε γραμμέ που είχαμε δώσει προ τα κράτη-μέλη σε μια απόπειρα να τις βοηθήσουμε να αξιολογήσουν την κείμενη νομοθεσία, διαπιστώσαμε ότι σε πάρα πολλέ περιπτώσει και στα ιατρικά επαγγέλματα τα κράτη-μέλη είχαν κάποιες δυσκολίες ε, ε, ή δεν ήταν πρόθυμοι ή δεν ακολούθησαν επακριβώς τι κατευθυντήριε γραμμέ που δώσαμε να εξηγήσουν τι είναι η δεν ηταν προθυμοι η δεν ακολουθησαν επακριβω τι κατευθυντηριε γραμμε που δωσαμε να εξηγησουν τι ειναι η αναλογικοτητα ε, και τι σχέση υπάρχει με την νομοθεσία του και κατά πόσον είναι είναι αναλογική νομοθεσία ή όχι. Αυτά βέβαια ε, ε, προέκυψαν και από μια πολύ διεξοδική ανάγνωση και εξήγηση από το δικαστήριο. Το δικαστήριο πολλές φορές έλεγξε την νομοθεσία περί αναλογικότητας και έγινε και στον τομέα της υγείας και μάλιστα πολύ συχνά. Ε, εξετάσαμε αυτέ τι υποθέσει πάρα πολύ προσεκτική και προσπαθήσαμε να δώσουμε τι απαραίτητε πληροφορίες στα κράτη-μέλη στα πλαίσια αυτή τη διαδικασία. Βέβαια δεν οδήγησε στα αποτελέσματα τα οποία ελπίζαμε και γι' αυτό τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει μια πρόταση προκειμένου να υπάρχει μια πιο διαρθρωμένη προσέγγιση ε, αλλά, και αυτό δεν αλλάζει και τα όσα έχουμε κάνει στα τομέα της αμοιβαία αξιολόγησης, βασίζεται στην ομολογία του δικαστηρίου. Θα δείτε λοιπόν ότι όσον αφορά την ουσία της πρότασης, ε, πρόκειται για αυτά τα οποία έχει αποφασίσει το δικαστήριο επανειλημμένος και όπως σας είπα και για τον τομέα της υγείας δεν επιβάλλει κάτι επιπλέον στα κράτη-μέλη, προσπαθεί να διευκρινίσει τι λέει το άρθρο 59 για την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα και η ίδια η συνθήκη, δηλαδή ότι η νομοθεσία θα πρέπει να είναι αναλογική για το στόχο που προσπαθεί να επιτύχει. Τι προσπαθούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη, πιέζοντά τα και λίγο, αφού είδαμε ότι οι κατευθυντήριε γραμμέ δεν έχουν και πολύ καλά αποτελέσματα, προσπαθούμε να βοηθήσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία υποτίθεται ότι θα κάνουν και βάσει τη ε, συνθήκη και βάσει του κείμενου παραγόγου δικαίου για τον τομέα ε, και τη υγεία. Αυτό σημαίνει περιττή γραφειοκρατία, Εμεί δεν το πιστεύουμε αυτό. Όλα τα κράτη-μέλη και κάποια το κάνουν σε, ήδη σε κάποιο βαθμό θα ε, ε, νομοθετήσουν λαμβάνοντα υπόψη για το κατά πόσον υπάρχει και... αναλογικότητα και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα το κάνουν αυτό με μια κοινή αντίληψη του τι ακριβώς γίνεται. Ε, πρέπει να δούμε λοιπόν και τι κάνουν τα κράτη-μέλη στα ε, πλαίσια της ίδιας διαδικασίας, όπως κάνετε και εσείς. Όταν καταρτίζετε νέα νομοθεσία, λαμβάνετε υπόψη κάποια στοιχεία, εφαρμόζετε τα κριτήρια και αξιολογείτε βάσει των κριτηρίων που έχει καθαρίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν υπάρχει λοιπόν περιττέρω επιβάρυνση και περαιτέρω γραφειοκρατία. Επίσης δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για τα ίδια τα επαγγέλματα. Αντιθέτω, είχαμε κάποιε καταγγελίε από επαγγελματίε που λένε ότι υπάρχει πολλή νομοθεσία και δυσχεραίνει τα πράγματα. Όχι. αυτό σημαίνει ότι ο νομοθέτης, ο ρυθμιστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία θα είναι σε αναλογική διάσταση και εν τέλει θα είναι προ όφελο των επαγγελματιών. Δεν δυσκολεύουμε λοιπόν τη ζωή στους επαγγελματίες, ίσα ίσα προσπαθούμε να τους διευκολύνουμε και να τους δώσουμε περισσότερο χρόνο για την πραγματική τους δουλειά, για αυτό που πρέπει να κάνουν, αντί να πρέπει να αντιμετωπίσουν γραφειοκρατία που ε, μπορεί να έχουν τα κράτη-μέλη ε, με αναλογικό τρόπο. Η πρόταση επίσης περιλαμβάνει και κάποιες δικλείδες ασφαλείας ή μάλλον δυνατότητες για τα κράτη-μέλη όπως ε, προβλέπουν και οι κανόνες και η νομολογία του δικαστηρίου για να έχουν το επίπεδο προστασίας που μπορούν να έχουν, να δουν κατά πόσον θέλουν να έχουν καλύτερη ρύθμιση. Όλα αυτά βέβαια στα πλαίσια της αναλογικότητας, αλλά όπως σας είπα αυτό είναι το σύνηθες και έτσι γίνεται ε, γενικότερα. Δεν προσπαθούμε λοιπόν να δυσκολέψουμε τη ζωή των κρατών μελών, δεν ε, προδικάζουμε το αποτέλεσμα, δεν περιγράφουμε πώς θα γίνονται οι ρυθμίσεις. Λέμε απλώς ότι όποτε σκέφτεστε να νομοθετήσετε, δείτε καλύτερα τι περιλαμβάνει νομοθεσία, εξετάστε την πλευρά της ανατολικότητας, εξετάστε τα κριτήρια τα οποία έχει αναπτύξει ε, το δικαστήριο για να εξηγήσει αυτά τα κριτήρια. Και τι σημαίνει αυτό συστηματικά για την αναλογικότητα. Και επίσης σας είπα μην θεωρήσετε ότι αυτό θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα για τα ιατρικά επαγγέλματα. Ε, θεωρούμε ότι καλή ιδέα θα ήταν να παραμείνουν και να καλύπτονται και από την οδηγία ε, και αν υπάρχουν κάποιες ιδιωτερότητες τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, είμαστε διατεθειμένοι να βελτιώσουμε το κείμενο προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Γκροστέτ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους για τις απόψεις που εξέφρασαν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο σύνολο των ερωτήσεων και των παρατηρήσεων που έγιναν, γιατί πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, μας επιτρέπει να διευκρινίσουμε τα σκοτεινά σημεία. Ε, πρόκειται για μια γνωμοδότηση την οποία υποβάλλουμε σε έκθεση της ΥΜΚΟ. Βεβαίως γνωρίζω τον εισηγήτη και έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί. Μπορώ να επιβεβαιώσω λοιπόν αυτό που έλεγε πριν από λίγο ο συνάδελφος Λίζε, ότι πράγματι ο κύριος Φαμπ έχει την ίδια θέση με αυτή που την δική μας, δηλαδή ότι πρέπει να εξαιρεθούν τα επαγγελμάτα του χώρου της υγείας. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και ε, επί μακρό χρονικό διάστημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έρχεται και ξανάρχεται. Το είπαν ορισμένοι συνάδελφοι που έλαβαν το λόγο ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τα επαγγέλματα του χώρου της υγείας σαν οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Δεν ε, μπορούμε να τα εξομοιώσουμε με την παροχή υπηρεσιών. Γιατί εδώ μιλάμε για την δημόσια υγεία, μιλάμε για επαγγέλματα στα οποία κάθε κράτος μέλος έχει νομοθεσία ελέγχου τους, ε, κατοχήρωσης τους και ελέγχου τους, επομένως δεν μπορούμε να τα δούμε σαν υπηρεσίες, παροχή υπηρεσιών. Επίσης, αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έρχεται και μας λέει ότι η πρότασή τη δεν θα αλλάξει τίποτα. Ε, αφού δεν θα αλλάξει τίποτα, γιατί υποβάλλεται πρόταση, τι νόημα έχει. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Εάν έρχεται μια πρόσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα αλλάξει κάτι στην υφιστάμενη κατάσταση και έχει προστιθέμενη αξία να το κάνουμε, διαφορετικά να μην το κάνουμε. Ε, είναι πολλά και διάφορα τα επαγγέλματα της υγείας, το είπαν και οι συνάδελφοι, καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών στην Ευρώπη. Επομένως, εάν τίποτα δεν θα αλλάξει, που μας λέει η Επιτροπή, γιατί να δημιουργήσουμε ανησυχία σε όλους αυτούς τους επαγγελματίες. Ε, ιδιαίτερα, μάλιστα, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη η ε, οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στο άρθρο 59 της οποίας ρυθμίζεται το ζήτημα αυτών των επαγγελμάτων. Αν κοιτάξουμε λοιπόν αυτό το άρθρο 59 δεν βλέπω τι περισσότερο προσθέτει η πρόταση της Επιτροπής. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω ότι θα δημιουργήσει επιπλέον γραφειοκρατία. Και για να το τεκμηριώσω αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στο ε, άρθρο 6 ε, της πρότασης. Προτείνει μια διαδικασία εξαιρετικά περίπλοκη γιατί θα έπρεπε να ε, αποδειχθεί ότι κληρούνται τα εξαιρετικά ε, περιοριστικά κριτήρια του άρθρου 6 και ζητώ από τους συναδέλφους που ε, ανησυχούν γι' αυτό να διαβάσουν τα κριτήρια του άρθρου 6. Η Επιτροπή πάλι μας λέει ότι δεν θα υπάρξουν επιπλέον διαδικασίε, ότι θα αξιοποιούμε τα υφιστάμενα κριτήρια. αυτό δεν πιστεύω ότι ισχύει, γιατί όταν ζητείται συστηματικός ε, έλεγχος αυτών των κριτηρίων, κάποιος οργανισμός θα πρέπει να τον ασκεί. Ο συνάδελφος ή συνάδελφος από την ΚΟΕ με εξέπληξε, γιατί στην πραγματικότητα μιλάει για περισσότερη φιλελευθερωποίηση του, του, του χώρου αυτού, για απορρίθμιση μάλλον του χώρου αυτού, ενώ αυτή τη στιγμή λειτουργεί σωστά. Όπως είπα, ο χώρος της υγείας δεν είναι ένας, ε, ε, μια αγορά υπηρεσιών, δεν πρόκειται για μια αγορά στην οποία η αύξηση του ανταγωνισμού θα μειώσει τις τιμές. Ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή στον τομέα της υγείας έχουμε τεράστια γραφειοκρατία. Μας το λένε οι γιατροί, οι επαγγελματίες του χώρου, ότι έχουμε να συμπληρώνουμε ατελείωτες ε, φόρμες και χαπιά και στοιχεία που μας ζητάνε τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε κάθε χώρα. Ελάτε λοιπόν στη θέση τους όταν υπάρχει ήδη αυτή η γραφειοκρατία. Λογικό δεν είναι να έχουν μία στάση επικριτική απέναντι σε αυτή την ε, πρόταση όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχει ήδη η αίσθηση και η εικόνα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το μόνο που κάνει είναι να προσθέτει γραφειοκρατία. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι έχουμε στην διάθεσή μας τα κράτη-μέλη μία η φυστάμενη νομοθεσία η οποία μας καλύπτει. Η Επιτροπή λέει εντάξει υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη νομοθεσία. Άρα τι κάνουμε για να ε, επιλύσουμε ορισμένες εξαιρέσεις, ορισμένα, ορισμένες περιπτώσεις όπου η νομοθεσία αυτή δεν έχει εφαρμοστεί σωστά στα κρατημέλη, δεν λειτουργεί σε κάποιο κράτος μέλος. Θα δημιουργήσουμε μια γενικότερη διαδικασία που θα δημιουργεί ε, γραφειοκρατικά εμπόδια. Δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ε, μεμονωμένα προβλήματα ελπίζω με τη συνεργασία όλων των συναδέλφων και με τη συνεργασία που θα έχουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά να καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε για το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 7 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας ΕΝΒΙ θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΙΜΚΟ έχει προγραμματιστεί για τις 20 ή 21 Νοεμβρίου του 2017. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης. Πρόθεση της χρήσης ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Άικχαουτ και θα του δώσω τον λόγο αυτής αμέσως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ε, ένα από τα θέματα του χειμερινού πακέτου που παρουσίασε η Επιτροπή ε, στα τέλη του έτους πρόκειται για μια μεγάλη δεσμή μέτρων που αφορά την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, σχεδιασμό, σχέδιο, design. Ε, και ε, η Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε θέματα ε, κριτηρίων βιωσιμότητας, βιοκαυσίμων και βιομάζας. Θα σταθώ σε αυτά εντός ολίγου, αλλά βεβαίως ως Επιτροπή Περιβάλλοντος πρώτα και κυριότερα θα πρέπει να εντρυφήσουμε στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα γνωμοδοτήσουμε για την Επιτροπή Ήτρε που είναι αρμόδια επί της Επιτροπή και κυρίως αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι υπέρ των ανανεώσιμων. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο του 20% για το 2020, τον οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα πετύχει, παρά το γεγονό ότι δεν θα τον πετύχει κάθε χώρα τον εθνικό τη στόχο. Κάποιε χώρε έχουν δυσκολίε, μεταξύ των οποίων και η δική μου, οι 100 χώρε. Βεβαίω, ε, το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από εκεί και πέρα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναγνωρίσουμε ότι η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020 ήταν ε, ε κομβική σημασία για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να σας πω και πάλι για τι κάτω χώρε. Εάν δεν υπήρχε η οδηγία για τι ανανεώσιμε, δεν θα υπήρχε συμφωνία για την ενέργεια στις κάτω χώρες, η οποία αυτή τη στιγμή ε, προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπετε λοιπόν ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προωθούνται σε κάθε χώρα λόγω της οδηγίας και του στόχου του 2020. Ο στόχος που για το 2020 σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ετήσια αύξηση της τάξης του 5% μέχρι το 2020. Εάν τηρήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 27%, αυτό σημαίνει ότι μετά το 2020 η αύξηση θα μειωθεί από το 5% ετησίως στο 1% ετήσια αύξηση μετά το 2020 ένα ποσοστό το οποίο μειώνεται παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνονται πιο, ανα... πιο ανταγωνιστικές και αυτή είναι μια επιλογή την οποία δεν θα μετανιώσουμε αν δούμε το μελλοντικό ενεργειακό προφίλ μας. Πρόκειται λοιπόν για μια κατεύθυνση την οποία σαφώ και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο το επίπεδο φιλοδοξία. Και επίση θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες και μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη από το ECOFES και το Τεχνικό Ινστιτούτο της Βιέννης, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από δύο εβδομάδες, που λέει ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο κάτω του 35% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσουν οι επενδύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανανεώσιμες θα σταματήσουν οι επενδύσεις. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι πηγαίνουμε αντίθετα σε αυτό το οποίο ισχυριζόταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούνκερ, ο οποίος ε, έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ο υπαριθμόν ένα ε, παράγον στις ανανεώσιμες. Αν θέλετε λοιπόν να είστε το ε, νούμερο ένα και απ' την άλλη μειωθούν οι επενδύσεις, κάτι δεν πάει καλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευτυχώ βεβαίω εμείς μπορούμε να τα διορθώσουμε, γιατί ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά θα αναφερθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2014. Ευτυχώ λοιπόν εμείς ως Κοινοβούλιο δεν χρειαζόμαστε να είμαστε οι υπάλληλοι του Συμβουλίου, είμαστε στο Κοινοβούλιο εδώ. Ε, η ίδια μελέτη από το Ινστιτούτο της Βιέννης και το ΕΚΟΦΕΣ λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα τα δικαιώματα των επενδυτών θα δοθούν και με στόχο 45%. Και αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί αν έχουμε και έναν ε, τελικό στόχο του 40%, ο οποίος προτείνεται και από τον εισηγητέ σας εδώ στην Επιτροπή ΕΜΒΗ. Αν δούμε λοιπόν το πακέτο, το πιο λογικό είναι να έχουμε 45% ενεργειακή απόδοση, 45% ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και αυτό φυσικά θα βοηθήσει και γι' αυτό και ο εισηγητή σα εδώ προτείνει 45%. Και θα ήθελα να δείτε τις μελέτες οι οποίες ε, ε, αποδεικνύουν ότι αυτά είναι τα κατάλληλα στοιχεία. Ε, μετά από εκεί και πέρα βέβαια θα υπάρξουν εθνικοί στόχοι. Είμαι βέβαιος ότι αυτή θα είναι μία από τις ουσιαστικές συζητήσεις στην Επιτροπή Ήτρε. Αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι χρειαζόμαστε εθνικούς στόχους προκειμένου να μπορέσουμε να ε, έχουμε καινοτομία σε κάθε κράτος μέλος. Περνάμε τώρα στα ανα... των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ε, ε, κριτηρίων βιωσιμότητα ε, μέσω βιομάζας. Πόσο χρόνο έχω κύριε Πρόεδρε, γιατί μου κάνετε νόημα. Ένα λεπτό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση κύριε Πρόεδρε. Άντε δύο. Δύο, ε. Καλά. δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει λοιπόν να τα πω πιο γρήγορα. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είχα λίγο περισσότερο χρόνο για το θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πιο πολύ χρόνο για το θέμα αυτό. Λοιπόν, για τη συζήτηση για τα βιοκαύσιμα πρώτη γενιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει σταδιακά να πάμε στο 3,8% και αυτό να είναι το ανώτατο για το 2030. Αποφάσισα αυτό να μην το αλλάξω. Αλλά πιστεύω ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, πολύ ομοί και ε, δεν κάνει διάκριση μεταξύ καλών και κακών, μεταξύ πρώτης γενιάς και δεύτερης γενιάς. Και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τα κριτήρια εδώ ως κριτήρια βιωσιμότητας. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι η Επιτροπή μας μόλις ενέκρινε την... Ε, έκθεση για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών που στη Συμβαστική πρόταση 20 λέμε ότι θέλουμε να έχουμε αυτή την αλλαγή της χρήσης γης. Και επομένως είναι αυτό το οποίο μόλις εγκρίναμε. Αν υπάρχει κάποιος λοιπόν ο οποίος έχει πρόβλημα με τη συγκεκριμένη αλλαγή, να ξέρετε ότι μόλις το εγκρίναμε και πρέπει να υπάρχει και συνέπεια. Και γιατί το Κοινοβούλιο επανειλημμένως έχει ζητήσει να εξαιρεθεί η χρήση του φινικελαίου για τα βιοκαύσιμα. Ε, ξέρετε ότι δεν μπορούμε ως κοινοβούλιο να πούμε ότι δεν θέλουμε το φινικέλο, γιατί αυτό θα, έχει, θα δημιουργήσει προβλήματα στον ΠΟΕ. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις του ΠΟΕ, επομένως μπορούμε να βελτιώσουμε καλύτερα τα κριτήρια, τα οποία θα οδηγήσουν ε, στην αφαίρεση τελικά του, καταλο... του φινικελαίου από τον κατάλογο. Αυτό είναι για τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει και περιθέριο για εθανόλη πρώτης γενιάς που θα αυξηθεί σε αυτό το ανώτατο όριο του 3,8%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει για όλα ε, τα βιοκαύσιμα τα οποία καλλιεργούνται και υπάρχει δυνατότητα για βιοκαύσιμα από καλλιέργειες τα οποία ε, θα πληρούν ε, τα κριτήρια και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις βιοθανόλης οι οποίες μας είναι γνωστές. Τώρα, για τα προηγμένα βιοκαύσιμα Πιστεύω ότι αν εξετάσουμε το μέλλον των μεταφορών θα πρέπει να υπάρχει και πιο δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας και βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει ε, ε, και μεγάλη συζήτηση και για ε, μεταφορά επιβατών αλλά και για εμπορεύματα. Θα υπάρχει μέλλον για τα βιοκαύσιμα ή θα περάσουμε στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Προτείνω λοιπόν να υπάρχει ο στόχος του 6,8%, να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ επιλογών ηλεκτρικής ενέργειας και επιλογών βιοκαυσίμων, ώστε να δείξουμε και σαφέστατα στους παραγωγούς προηγμένων βιοκαυσίμων και εδώ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την αεροπορία, διότι εκεί θα πρέπει να στραφούν κυρίως τα βιοκαύσιμα προηγμένης γενιάς, μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο και αν περιλαφθεί και η αεροπορία σε αυτό το τομέα, όντως θα, προ... θα είμαστε ε, στα ημεία. Ξέρετε ότι υπάρχει το περιβόητο παράρτημα 9, το οποίο ε, είναι αντικείμενο επικρίσεων και από τον διατροφικό τομέα και από άλλους που λένε ότι χρησιμοποιούμε κάποιες από αυτές τις ενώσεις, τις χρησιμοποιούμε στις χημικές μας εφαρμογές και τώρα περιλαμβάνονται στο, άρθρο, στο παράρτημα 9 και θεωρούνται προηγμένα βιοκαύσιμα. Υπάρχει λοιπόν ανταγωνισμός και εγώ προτείνω να συμπεριλάβουμε και τα κριτήρια για τις εκπομπές, τα οποία θα μας δείξουν ότι αυτά τα οποία εφαρμόζονται και σε χημικό επίπεδο που ε, είναι υψηλότερη χρήση, τότε τα ενδιάμεσα κριτήρια εκπομπών θα εξασφαλίσουν ότι δεν χρησιμοποιούμε λανθασμένες ενώσεις για προηγμένα ε, βιοκαύσιμα. Ε, υπάρχουν λοιπόν μεγάλες συζητήσει για διάφορες ε, χημικές ουσίες και για τα χημικά. Και να ολοκληρώσω γιατί έχω και τη βιομάζα. Και εδώ είναι πολύ ισχνή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δείτε τι γίνεται εκεί, υπάρχει κάτι το οποίο είναι σίγουρο. Για παράδειγμα, οι εισαγωγέ ε, πάλετ για χρήση βιομάζας από Ηνωμένε Πολιτείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποκλείονται. Αν δείτε την αξιολόγηση επιπτώσεων, υπάρχει λόγος να πούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, τα απορρίμματα και τα κατάλοιπα και αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη βιομάζα και θα έχουμε ε, και τους στόχους μας και αυτοί που λένε ότι δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Αν δείτε τα απορρίμματα και τα κατάλοιπα, έχουμε 50%. Να χρησιμοποιούμε λοιπόν τα κατάλληλα υλικά και για τη βιομάζα και αυτό προτείνω στην έκθεσή μου. Χρειάστηκε να συντομεύσω λίγο, αλλά τέλος πάντων δεν θα πω άλλο. Σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι είναι ενδιαφέρουσα πολύ αυτή η συζήτηση, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα τη Επιτροπή. Να δώσω το λόγο τώρα στου συζητητέ στο σκεύο του ΕΛΚ. Καταρχάς, την κυρία Πετήρ. Τέσσερα λεπτά, παρακαλώ, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη Συμφωνία των Παρισίων και βάσει και των ευρωπαϊκών στόχων ενεργειακής πολιτικής και προστασίας του κλίματος, πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν κοινό στόχο όσον αφορά το ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική ενεργειακή κατανόληση ε, μέχρι το 2030. Αλλά ο στόχος αυτός θα πρέπει να είναι και ρεαλιστικός. Κατά την άποψή μου, η μείωση του ποσοστό των συμβατικών καυσίμων αποστέλει λανθασμένο μήνυμα στους πιθανούς επενδυτές. Η τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν ε, την ποσόστοση χρήσης ε, βιοκαυσίμων και να παραμείνει στο 7% μέχρι το 2030 και για να μετριάσουμε και τις αρνητικές συνέπειες ε, της άμεσης χρήσης γης, Στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να καταλήξουμε ε, στο στόχο στον οποίο θέλουμε να φτάσουμε και για οδικές ε, και για σιδηροδρομικές μεταφοράς ε, και θα αφορά και όλα τα καύσιμα μέχρι το 2030. Οι στόχοι εν γέννη θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξοι από αυτούς που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν αναφερόμαστε στην ε, μεικτή κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020 και από το 2021 και μετά, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες ε, του κάθε κράτους μέλους, θα πρέπει να υπάρχει και ε, περιθώριο να αποφασίζουν για τα ποσοστά για τη χρήση καυσίμων και υγρών βιοκαυσίμων. Αυτό περιλαμβάνει και καύσιμα από βιομάζα. Και φυσικά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η έμεση ε, αλλαγή χρήσης γης. Κατά την άποψή μου, πρέπει να υπάρχει μια παρέκκληση από τα όρια τα οποία συζητούμε τώρα. Εισάγεται το 60% των ζωοτροφών Πρόκειται ε, για προϊόντα γενετικώς τροποποιημένα, τα οποία δεν θα θέλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εναλλακτική λύση θα ήταν να ε, χρησιμοποιούν αυτά για παραγωγή καυσίμων, τα οποία θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε ε, με αυτή την παραγωγή. Εγώ υποστηρίζω τα κριτήρια βιωσιμότητας για τη βιομάζα, για αυτές τις καλλιέργειες, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον γραφειοκρατικό άχθος και τα όρια δεν θα πρέπει να καθορίζονται βάση... Ε, συγκεκριμένου καυσίμου, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και όλη την έκταση βιομάζας. Επειδή ε, οι καλλιέργειες αυτές δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά στοιχεία διαχείρισης των ζασών από τους ιδιοκτήτες. Πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση η οποία θα πρέπει να βασίζεται στους κείμενους κανόνες και θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται βάσει πρωτοβουλίας των κρατών μελών. Θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Γιώ Λάινεν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον κύριο Άικχαουτ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και θα έπρεπε να έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι και πολύ περίπλοκο. Και θα πρέπει να δούμε προς τα που οδεύουμε και που θα φτάσουμε. Για το σημείο κίνηση. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι οι στόχοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ χαμηλοί. 27%, 72% συγγνώμη, μέχρι το 2030 είναι business as usual. Δεν α, στέλνει αυτό οποιοδήποτε σαφέ μήνυμα προ του εμπλεκόμενου φορεί, την οικονομία, την κοινωνία. Θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά οι στόχοι αυτοί. Τώρα πόσο θα πρέπει να, να αυξηθούν, αυτό δεν θα μα βρει σύμφωνος ενδεχομένω όλου μετά τη Συμφωνία του Παρισίου έχουμε πει ότι για να πετύχουμε τους στόχους που θέσαμε εκεί θα πρέπει μέχρι το 2030 να πετύχουμε 40%. Βέβαια, ο καθένα μπορεί να βρει ό,τι έρευνα και μελέτη θέλει για να υποστηρίξει σε ποιο σκοπό θέλει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε το, 40, να ξεπεράσουμε το στόχο αυτό και να ταχθούμε προ το 40% για το 2020 τώρα. Είχαμε εθνικά δεσμευτικού στόχους. Γιατί η όσο υπάρχει μεγάλη διαφορά. Οι μεν δεν κάνουν τίποτα και οι άλλοι αγωνίζονται και τρέχουν. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν δεσμευτικοί στόχοι ανά κράτος. Επίσης, καλό στην πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ενίσχυση του καταναλωτή. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε παραγωγοί και καταναλωτέ για ίδια χρήση δηλαδή στον τομέα αυτό των ε, ανανεώσιμων. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν αυτή την παραγωγή ιδέα ενέργεια. Επίση να τοποθετηθώ για την θέρμανση και την ψήξη. Θα πρέπει να αυξηθούν, θεωρώ, τα ποσοστά της χρήσης ανανεώσιμων ενεργειών. Η βιομάζα θα διδραματίσει ασφαλώς ρόλο αλλά όπως ε, ξέρετε χρειαζόμαστε και κριτήρια βιωσιμότητας. Δεν μπορούμε να έχουμε τη βιομάζα και να χρησιμοποιείται στον τομέα της θέρμανσης χωρίς περαιτέρω σκέψη. Τώρα για τα βιοκαύσιμα. Πριν από 15 χρόνια υπήρχε μεγάλη μόδα για τα βιοκαύσιμα. Τότε ήταν μόδα. Τώρα είναι ο δαίμονας αυτό. Και τα κατηγορούμε. Για τα βιοκάψιμα. θεωρώ ότι θα πρέπει να θέσουμε κριτήρια, κριτήρια βιωσιμότητας. Θα πρέπει να συμβάλλουν στην ε, προστασία του κλίματος και εδώ θα πρέπει να κάτσουμε να κοιτάξουμε με προσοχή τους καλούς και τους κακούς από την πρώτη στη δεύτερη γενιά αλλά και εντός της πρώτης γενιάς. Όλες οι μελέτες καταδεικνύουν ότι τα βιοκαύσιμα, το φινικέλαιο και η σόγια είναι χειρότερα και σε ό,τι αφορά την εθανόλη. Υπάρχουν ε, φυτά τα οποία δεν είναι αρνητικά, είναι ουδέτερα. Μην σας πω ότι σε μερικές περιπτώσεις είναι και θετικά. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι θα πρέπει να ορίσουμε τις προτάσεις μας. Ο εισηγητής αναφέρει και ενισχύει τα κριτήρια αποδοτικότητας και τα κριτήρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας. Εμείς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μέχρι το 2025 ε, αποσυρώμεθα. Μπορεί να τα κάνουμε όλα τόσο αυστηρά, αλλά μετά το 2025 δεν θα έχουμε τίποτε πλέον. Θεωρώ ότι αυτό ξεπερνάει το στόχο μας για τη βιομάζα. Να συμφωνήσω σε ό,τι αφορά Θα πρέπει να εξελιχθούν τα θέματα της ε, μελάσας και των ελαίων, αλλά το θέμα είναι αν όλες οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές για πολλά μεγαβάτ, μήπως αυτό είναι υπερβολικό ε, και η Κομισιόν συστήνει 20 ΜΒ, εγώ θα σύστηνα μάλλον 5 ΜΒ, γιατί πραγματικά οι εγκαταστάσεις μας ανησυχούν. Είναι 300 στον αριθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από 20 ΜΒ. Και πιστεύω ότι στην περίπτωση αυτή θα έρθουν από, τα Ηνωμένα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το πνεύμα θα ακολουθήσουν και οι τροπολογίε μα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει και Πρόεδρο. Επόμενο ομιλητή από το ECR, η κυρία Βυσνιευσκά. Σας ευχαριστώ πολύ. συνάδελφοι, πιστεύω ότι το προσχέδιο που έχουμε μπροστά μας, ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι υπερβολικά φιλόδοξο, θα το έλεγα. Δηλαδή, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω αυτό με κάποιες παρατηρήσεις που έχω να κάνω. Ο εισηγητής κάνει κάτι που δεν συνηθίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή να προτείνει έναν στόχο εξαιρετικά υψηλό, τον οποίο γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να πετύχουμε, γιατί δεν πρόκειται να το επιτρέψουν αυτό τα κρατή-μέλη. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το περσινό, θέτει ένα στόχο της τάξης του 30%, ενώ η εισηγητής προτείνει 45%. Ε, επιπλέον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους ε, εθνικούς στόχους ένα άλλο ζήτημα ευαίσθητο που προκαλεί δυσκολίες και το βλέπουμε σε ολόκληρη την ε, έκθεση είναι το ζήτημα των βιοκαυσίμων που παράγονται από καλλιέργειες και από τη δασοπονία και επίσης το ζήτημα των απολειών. Ε, συγγνώμη, το, το ζήτημα της παραγωγής από απορρίμματα. Ισχύει πράγματι ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε περισσότερα, περισσότερο και πιο αποτελεσματικά αυτές τις πηγές βιοενέργειας. Όμως, όπως διαβάζω εγώ το προσχέδιο της εκθέσης, μετά το 2020 η παραγωγή ε, βιοενέργειας από τον γεωργικό τομέα ε, και, και με τέτοιες μεθόδους θα αποκλειστεί πλήρως. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Επίσης λέγεται ότι από το 2021 και μετά θα πρέπει να πάψει η υποστήριξη, η ενίσχυση που δίνεται στα προγράμματα παραγωγής ενέργειας από τα αστικά απορρίμματα. Αυτό πιστεύω ότι δεν είναι σωστό, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ε, σε πολλές περιοχές της Ευρώπης ε, χιτά, όπου τα απορρίμματα καίγονται. Και παρόλο που αυτό δεν είναι ε, σε καμία περίπτωση ο πιο αποτελεσματικό τρόπο παραγωγή ενέργεια, το αντιλαμβάνομαι αυτό, δεν θα είναι δυνατόν μέχρι το 2021 να καταφέρουμε να κλείσουμε όλε αυτέ τι μονάδε. Άρα πιστεύω ότι θα έπρεπε καλύτερα να, να, θέσουμε πιο ρεαλιστικού στόχου εδώ. Η τροπολογία 36 πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση, ζητώντας τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν μια σειρά παραγωγή μεθόδων στι οποίε θα περιλαμβάνεται και η γεωθερμική. Αυτό το καλωσορίζω. Θα υποβάλω διάφορε τροπολογίε ε, για τα προβλήματα που σα ανέφερα, ιδίω εστιάζοντα στο ζητήματα των βιοκαυσίμων. Ο κύριο Χάτεμα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ε, εκπροσωπώ τον να ευχαριστήσω καταρχά τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανα και επίση ε, ο σκιώδης μα θα ήθελε να συμφωνήσει ότι η αύξηση τη φιλοδοξία των τομέα των νεώσιμων είναι απαραίτητη αν θέλουμε να πετύχουμε του στόχου μα ε, για την αλλαγή του κλίματος. Ε, εμείς πάντα ζητούσαμε 30% μέχρι το μέχρι το 2030. Οτιδήποτε κάτω από αυτό δεν θα το δεχτούμε. Και για να υπάρχει νομισματική βεβαιότητα και να τονωθούν οι επενδύσεις και οι τεχνολογικές ε, εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να υποστηρίξω την ε, πρόθεση των επιπέδων αυτών σε ό,τι αφορά τις μεταφοράς μου προκαλεί έκπληξη αλλά και φρίκη το αίσθημα τεζαβού που έχω. Δεν είναι, το έχω γράψει εγώ το κείμενο, σας το λέω. Τα ερωτήματα λοιπόν που τίθενται για τα βιοκαύσιμα της πρώτης γενιάς και τα προηγμένα βιοκαύσιμα, τα κριτήρια βιωσιμότητας μου θυμίζουν αυτά που χρησιμοποιήσαμε και πριν από μία δεκαετία και για την οδηγία για το άλλο. Θεωρώ ότι γενικά πρέπει να αλλάξουμε επιτέλους ε, τροπάρι για τα θέματα αυτά και να γυρίσουμε τη σελίδα σε ό,τι αφορά την ε, δυνατότητα των βιοκαυσίμων πρώτη γενιά και τη δυνατότητα αλλαγή τη τάση μα, αυτό έχει τρομολογηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σταδιακή μείωση λοιπόν των βιοκαυσίμων που βασίζονται σε Σπαρτά. Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των βιοκαυσίμων, πρέπει να σα πω ότι και το παράρτημα 9 και το σύστημα πολλαπλή καταμέτρηση με ενοχλεί. Αν δεν θέλουμε κάθε 2, 3, 4, 5 χρόνια να κάνουμε την ίδια συζήτηση, που πιστεύω ότι θα έπρεπε. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι. Η αλλαγή της πορείας μας ε, συνολικά φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολη και οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να συνοδευτεί από καθοδήγηση. Γι' αυτό αυτή τη φορά εστιαστήκαμε πολύ στην μείωση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα βρει σύμφωνο όλο το Κοινοβούλιο. Ωστόσο, τι σημαίνει αυτό στην πράξη κατά πόσον θα λάβουμε υπόψη τον έλεγχο ή όχι. Αυτό θα πω είναι ένα από τα βασικά ζητήματα στις πολιτικές ομάδε, μεταξύ των οποίων και στη δικιά μου. Uh, Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητή από το EFTD, ο κ. Ακούτε μουσική από κάπου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς προφανώς και είμαστε υπέρ ε, της έκθεσης του συναδέλφου Άικχουτ Eichhout, διότι πιστεύουμε πραγματικά στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για να επιτευχθούν όμως αυτή η φιλόδοξοι στέχη, δεν υπάρχει χώρος για τα ορυκτά καύσιμα, ακόμα και αν προέρχονται από τα απόβλητα. Και επίσης θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας χώρος για την καύση των αποβλήπτων, που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρείται μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ της οποιασδήποτε ενίσχυσης για τα ορυκτά καύσιμα και οποιοδήποτε ε, ενίσχυση και κίνητρο για την καύση των αποβλήτων. Είναι αντίθετα με όλη αυτή την ιδέα της κυκλικής οικονομίας που προσπαθεί να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα πρέπει να προωθήσουμε την ηλιακή, την αιωλική ενέργεια, να δώσουμε έμφαση στην ενεργειακή εξοικονόμηση και να βοηθήσουμε για την ε, καλύτερη ε, χρήση ενέργειας από τις μεταφορές. Και στην βιομηχανική μπορούμε να έχουμε αλλά, ε, κάποια πρόοδο, αλλά μόνο αν την περιορίσουμε στα απόβλητα, ε, στα κατάλοιπα και σε άλλα επεξεργασμένα τα προϊόντα που δεν μπορούν να έχουν άλλη εναλλακτική χρήση. Γι' αυτό το λόγο ο κατάλογος των υλικών που χρησιμοποιούνται για τα προηγμένα βιοκαύσιμα που είναι στο παράρτημα 9 μας δημιουργεί ακόμα κάποιες αμφιβολίες, ιδίως για τις πρώτες ύλες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για άλλους βιομηχανικούς σκοπούς πριν γίνουν καύσιμα. Θεωρούμε ε, ότι θα πρέπει να υπάρχει η αρχή της ε, βαθμιδών χρήσης των πόρων και επίσης θεωρούμε ότι τα παραδοσιακά βιοκαύσιμα, ο παράγοντας Άιλουκ θα πρέπει να υπολογίζεται στις εκπομπές ε, των καυσίμων. Θεωρούμε ότι η επίτευξη αυτών των φιλοδοξιών θα είναι σίγουρα δύσκολη, παρά το γεγονός ότι συμφωνούν αρκεί από εσά, παρά το γεγονό ότι είναι, διότι είναι πολύ ισχυρό ακόμα το λόμπι των ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να πιέσουμε όμως για δεσμευτικούς στόχους για κάθε χώρα για τουλάχιστον 45% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030 και επίσης θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία η οποία θα βασίζεται πλήρως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2040. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Δύο λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Μπάλτσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιληφθεί ότι το 27% μέχρι το 2030 δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει επεξεργασία του στόχου αυτού. Συμφωνώ. Το ΕΛΚ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το 30% και τώρα ο εισηγητή ε, προτείνει παραπάνω ποσοστό. Είμαστε βουλευτέ και αποφασίζουμε τι θέλουμε. Δίκιο έχετε, αλλά καλό θα ήταν αν αυτή η στόχη ήταν και ρεαλιστική παράλληλα. Υλοποιήσιμη. Για τι ανανεώσιμε ενέργειε αναφέρουμε ότι μπορούν να δημιουργηθούν ε, θέσει απασχόληση ε, προωθείται η οικονομία, η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια δίνουν μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι η πυρηνική ενέργεια. Και κυρίως πρέπει να χρησιμοποιούνται και καθαρές πηγές ενέργειας δεδομένης της αλλαγή του κλίματος. Να ρωτήσουμε ποιος πληρώνει τελικά αυτή τη νέα μορφή ενέργειας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπε ότι ο στόχος είναι 27% μέχρι 2030. Αυτό συνεπάγεται διπλάσιο κόστος από το προβλεπόμενο. Μιλάμε για τεράστια ποσά τα οποία πρέπει να επενδυθούν και αυτό αποτελεί μεγάλη επιβάρυνση. Στην Επιτροπή αυτή μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σαν να είναι νύφη, που θέλουν να όλοι καλά σχόλια και κοπλημένα στο γάμο. Όλα καλά και ωραία αυτά. Αλλά τελικά συνεπάγονται τόσο μεγάλη επιβάρυνση για τα κάτι μέλη, που δεν είναι υλοποιήσιμη η στόχη αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια απόχρωση σε όλα αυτά, σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση τη Επιτροπής. ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Βλέπω ότι πολλοί επιθυμούν και υπάρχει μια σχετική πίεση να αλλάξει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πράγματι, ο ε, εισηγητής προσπαθεί να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, πιστεύω ότι τα εργαλεία που τελικά επιλέγουμε μάλλον θα δυσχεράνουν την προσπάθεια της Ένωση να επιτύχει τους στόχους της για την κλιματική αλλαγή. Ε, τα κριτήρια βιωσιμότητας για τις ΑΠΕ είναι ίσως υπερβολικά σε ορισμένες περιπτώσεις. το ίδιο και ο τελικός στόχος του 45%, δηλαδή του 45% της ενέργειας να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, που είναι 15% περισσότερο από τον αρχικό στόχο πρόταση της Επιτροπής. Καλό είναι καλή να θέτει φιλόδοξους στόχους, αλλά θα πρέπει κατά την άποψή μου να εξετάσουμε όλε τι επιλογέ ανανεώσιμων πηγών που έχουν στη διάθεσή μα, συμπεριλαμβανομένων και των βιοκαυσίμων, που μπορούν να συνεισφέρουν εάν χρησιμοποιηθούν σωστά είναι ανησυχητικό να έχουμε μια υπεραπλουστευμένη ε, ερμηνεία της έννοιας της βιωσιμότητας η οποία τελικά να μας περιορίζει, να μην μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε όσο θα έπρεπε στο μέλλον τα βιοκαύσιμα, ιδιαίτερα τα βιοκαύσιμα νέας γενιάς, των οποίων η χρήση αυξάνεται και τα οποία επιτρέπουν τα βιοκαύσιμα νέας γενιάς να μειωθεί σημαντικά η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Ε, έτσι κι αλλιώ ε, τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς σταδιακά θα σταματήσει η χρήση τους. Δεν θα μπορούσε να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη αυτό. Πρέπει να ενισχύσουμε, να ενθαρρύνουμε την έρευνα και την κοινοτομία έτσι ώστε να αναπτυχθούν βιοκαύσιμα νέας γενιάς πιο αποτελεσματικά. Στην Φιλανδία, από όπου κατάγομαι, Ένας από τους στόχους που μας δυσκολεύει είναι ακριβώς αυτός γιατί αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε ορισμένα καύσιμα που δεν θα καλύπτονταν από τα κριτήρια βιωσιμότητας για να πετύχουμε τους στόχους μας, τους κλιματικούς. Ε, ε, είναι λογικό αυτό αν λάβετε υπόψη σας και τη σημασία που έχει η δασοπονία για τη χώρα μου. Πρέπει λοιπόν πιστεύω να έχουμε μια ευρύτερη αντίληψη της χρήσης των βιοκαυσίμων για την επιτεύξη των στόχων. Οι λύσεις που θα βρούμε θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να βασίζονται σε μια ανάλυση του κατά πόσο είναι αποτελεσματική στην αγορά. Ελπίζω τελικά να βρούμε μια σωστή ισορροπία στις προτάσεις μας. Σας ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής, κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, πρωτού γίνει Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να καταστεί ηγετική δύναμη στις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και προσωπικά πρέπει να σας πω ότι όταν είδα την πρόταση του α, Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τελικά απογοητεύτηκα γιατί 27% δεν αντικατέχεται και από ιδιαίτερο επίπεδο φιλοδοξίας και αυτό που με απογοήτευσε ιδιαίτερως είναι το πλαίσιο με το οποίο υποτίθεται ότι θα πετύχουμε αυτό το 27% δεν είναι και πολύ καλά προκαθορισμένο το πλαίσιο αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να την επεξεργαστούμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προσεγγίσει κάπως πιο καλύτερα το όραμα του Ζαν Κλοντ Juncker. Από την άλλη, θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστέ στην προσέγγιση μα. και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σα πω ότι δυστυχώ τι προτάσει του Μπας Άικατ δεν μπορώ να τι προ... να τις ε, υποστηρίξω προσωπικά. 45% δεν είναι στόχο ε, ρεαλιστικός και υλοποιήσιμο. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι αυτό θετικό, αλλά πολύ απλά πιστεύω ότι δεν θα προκύψουν δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι. Και να μην ξεχνάμε και το εξή. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, γιατί και εγώ θέλω πιο υψηλού σκοπού ή στόχου. Οι ανανεώσιμε ενέργειε και αυτέ έχουν τα προβλήματά του. Τώρα δεν χρειάζεται εδώ πέρα να σα πω τα τη βιομάζα, όλα αυτά έχουν καταστεί σαφή. Και βλέπουμε και αυτό που προτείνει ο Μπά με επικριτικό πνεύμα. Μπά, να σου πω ότι γίνονται όλο και πιο πολλές συζητήσεις για την αιωλική ενέργεια. Δεν υπάρχουν αυτά σε απεριόριστο βαθμό. Θα πρέπει να υπάρξει και μία να, να, καταλάβουμε ότι υπάρχει και το ανταγωνισμό. Άρα, να βρούμε μία ενδιάμεση λύση ρεαλιστική. Το Συμβούλιο μας μιλά για έναν σταθερό σκοπό, για έναν διάδρομο. Ε, Δυστυχώ κάποιοι λένε ότι αυτό ο διάδρομο μπορεί να είναι και κάτω από 27% όχι. Ε, αυτή ήταν η πρώτη μου έκκληση. Αν μιλάμε για διάδρομο, θα πρέπει το κατώτατο όριο να είναι 27% και το ανώτατο να είναι και πάνω από το 30%. το 33% ενδεχομένω το οποίο είναι αποδοτικό σε ό,τι αφορά το κόστο. Αλλά βασικά θα πρέπει να δούμε πώ θα πετύχουμε το στόχο αυτό. Θα πρέπει να είναι σαφέ το τι θα συμβεί, αν τελικά κινδυνεύουμε να χάσουμε το στόχο μα. Και πολύ σαφέ είναι ότι τα κρατημέλη που κάνουν μεγαλύτερε προσπάθειε δεν θα πρέπει να τιμωρούνται τελικά. Χρειαζόμαστε λοιπόν benchmarks. Αν δεν υπάρχουν δηλαδή δεσμευτικοί στόχοι, τουλάχιστον να υπάρχουν αυτά τα benchmarks, αυτά τα ορόσημα βάσει των οποίων θα προσανατολιστεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρο. Επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι στην παρούσα φάση η τοποθέτησή μας ξεκαθαρίζει και πάει. Είμαστε διχασμένοι μεταξύ των φιλοδοξιών μας και της πραγματικότητάς μας πάντα. Και πιστεύω ότι αυτό που προτείνει ο Μπάς Άικχαουτ, το 45% θα πρέπει να προσαρμοστεί ελαφρώς προκειμένου να βρούμε μια τόπο, να πετύχουμε μια συμφωνία, εν περιπτώσει, και νομίζω ότι ο κύριος Πίτερ Λίζε είναι πολύ λογικός. Θα πρέπει να βρούμε ένα ελάχιστο επίπεδο το οποίο α, να το κατοχυρώσουμε, αλλά να προωθήσουμε και κάποιο άνωτατο όριο για τα κράτη-μέλη που θέλουν να το πετύχουν. Αυτό λοιπόν ήταν η πρώτη παρατηρήσή μου. Για την πρώτη γενιά, χαίρομαι αυτά που λέει ο κύριο Μπασάκη, που λέει ότι θα πρέπει να γίνει μια διάκριση σε ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς που επηρεάζουν. Αυτά που επηρεάζουν τον άλλο και αυτά που τα επηρεάζουν. Τα ευρωπαϊκά βιοκαύσιμα θεωρώ ότι ως πλήστον πληρούν τους όρους αυτούς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το βιοδίζελ και τη βιοεθανόλη. Και γιατί δεν τονίζω αυτό ιδιαίτερος. Γιατί οι πληροφορίες αυτές που αναφέρουν ότι μειώνουμε τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς αποτελεί ένα δείγμα και ένα μήνυμα προς την, στον κλάδο ότι αποσυρώμεθα ήδη. Ξέρουμε ποιες είναι οι, ποιο είναι το επίπεδο παραγωγής μας. 80% είναι σπαρτά για τρόφιμα. Μιλάμε για ζαχαρότευσλα και σε ό,τι αφορά άλλες πηγές βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς. Ε, με ικανοποιεί λοιπόν αυτή η λιγότερο περιοριστική στάση του εισηγητή, ο οποίος ε, διαχωρίζει το φινικέλαιο από τα ευρωπαϊκά σπαρτά. Αυτό θεωρώ ότι είναι θετικό και θα το κρίνουμε θετικά. Κατά δεύτερον, να θυμόμαστε ότι η παραγωγή των βιοκαυσίμων από το έλαιο, από, το, από την κραμβή, σημαίνει ότι παράγουμε και ζωοτροφές με πρωτεΐνη. Δεν θέλουμε να εισάγουμε στην Ευρώπη γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές και για κάθε τόνο λοιπόν έχουμε 600 κιλά βιοντίζελ και πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, χάρη στις οποίες δεν υποχρεούμαστε να εισάγουμε γενετικώς τροποποιημένα τροποποιημένη σόγια. Τελευταίο ζήτημα τώρα. Το θέμα της συμπερίληψης του τομέα της ε, αεροπλοείας σε ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα. Να δούμε τι γίνεται και στην ε, αμερικανική αγορά στη ΣΥΠΑ όπου είναι δεθμένοι να χρησιμοποιήσουν βιοκάψιμα ακόμα και στο στρατό. Πρέπει να έχουμε λοιπόν διαφορετική προσέγγιση. Και τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε τους καταναλωτές που μπορεί να είναι και παραγωγή. Αυτό θεωρώ ότι είναι για την διαφοροποίηση της παραγωγής και πιστεύω ότι θα έδινε ένα έναυσμα στους καταναλωτές να ενδιαφερθούν για τις νέες αυτές εγκαταστάσεις, το οποίο είναι θετικό για μας. Η κυρία Ντάλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επαναχωρήσει για το στόχο του 2020 για φιλόδοξους στόχους για τα βιοκαύσιμα και τις μεταφορές. Εάν θέλουμε να ανταποκριθούμε στους στόχους του COP21, θέλουμε να επιτύχουμε το συνολικό στόχο της ε, ε, διακοπής της χρήσης άνθρακα και τη μείωση των ε, αερίων θερμοκηπίου για τα και να πετύχουμε και τους στόχους για το 2030. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία θα ήθελα να σταθώ και θα ήθελα να τα θέσω διότι θεωρώ ότι είναι ουσιαστικά. Πρώτον και κυριότερον, η ανάγκη να υπάρχει δεσμευτικό στόχος για τα ανανεώσιμα πηγές ε, ενέργειας ε, στις μεταφορές για το 2030. Εγώ θα ήθελα οι αεροπορικές μεταφορές να συμπεριληφθούν ε, στο στόχο αυτό. Και επίσης ε, μαζί με αυτό θα πρέπει να αυξηθεί διαφάνεια για τον τύπο των βιοκαυσίμων που παρέχονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εθνικό επίπεδο, κάτι το οποίο ακόμα δεν υπάρχει ως πάγια πρακτική. Συμφωνώ πολύ τους ότι θα πρέπει να υπάρχει απαγόρευση για τη χρήση φενικελαίου ή τουλάχιστον να υπάρχει μία οριστική καταληκτική ημερομηνία για τη χρήση φινικελαίου για παραγωγή βιοδίζελ. Και επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε ε, τα προηγμένα βιοκαύσιμα και μάλιστα με σθένος, διότι αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην ε, ε εξάλληψη της χρήσης άνθρακα, εάν ξεκινήσουμε ευθύ εξ αρχής με αυτούς τους στόχους. Όσον αφορά τα προϊόντα των βιοκαυσίμων, θα πρέπει να είναι βιώσιμα και για τις αγορές θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ε, είναι βιώσιμα και αξιόπιστα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κάποια στοιχεία για τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Επίσης, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, ε, ακριβή ορισμό για τα βιοκαύσιμα, αντί να αποφασίσουμε για ένα κλειστό κατάλογο τώρα στο παράδειγμα 9α, ώστε να υπάρχει περιθώριο και για νέε τεχνολογίε στο μέλλον που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην αγορά. Κάτι σημαντικό επίσης είναι η ανάγκη να τονίσουμε και την ε, ηλεκτροκίνηση, αναφέρομαι στους στόχους του 2030. Δεν αρκεί απλώς να πούμε ε, ότι στις καθαρές μεταφορές πρέπει να έχουμε ε, βιοκαύσιμα, θα πρέπει να υπάρχει και ηλεκτροκίνηση, διότι θα μας βοηθήσει και αυτή σε αυτό το τομέα, ιδίω ε, για την επίτευξη υψηλότερων στόχων για το 2030. Θεωρώ ότι η ηλεκτροκίνηση είναι το πιο καθαρό καύσιμο το οποίο είναι διαθέσιμο και για τις ε, μεταφορές επιβατών, λοιπόν για τα ελαφρά οχήματα αυτό είναι το μέλλον. Πρέπει να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση στι μεταφορές και συμφωνώ εδώ και με την προσέγγιση του εισηγητή ότι θα πρέπει να υπάρχει ισχυρό πολλαπλασιαστικό παράγον για την ηλεκτροκίνηση, αλλά δεν ε, ε, αποκλείω και ένα στόχο για την ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για να επιτύχουμε το στόχο της ηλεκτροκίνησης. Βεβαίως ε, δεν ισχύει αυτό για την αεροπορία και την ναυτιλία και τα βαρέα οχήματα. Αυτή είναι τομεί στου οποίου πρέπει να βασιστούμε περισσότερο στα βιοκαύσιμα στο μέλλον και βεβαίω ε, για βιοκαύσιμα τα οποία θα είναι αποδεδεχμένα ότι παρήχθησαν με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην Κομισιόν τώρα. Την κυρία Μάρκες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Με χαρά ακούσαμε σήμερα το γεγονός ότι η Επιτροπή σας αναγνωρίζει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η δέσμευση για αυτή την νομοθεσία είναι σημαντικό, όπως ακούστηκε, όχι μόνο για την επίτευξη του στόχου να είμαστε παγκοσμίω ε, ηγέτης στην ανανεώσιμη πηγή, ε, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και για να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να επιτύχουν συλλογικά υψηλότερα ποσοστά χρήσης ΑΠΕ και ε, για μας αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 27% με αποτελεσματικό τρόπο και ως προς το κόστος. Όσον αφορά τους διάφορους μορφές που προτείνονται από την οδηγία, ε, η Επιτροπή θέλει να προωθήσει την ε, εξάλληψη της χρήσης άνθρακα και προτείνει επίσης να ενισχύσει το ε, πλαίσιο βιωσιμότητας. Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω εδώ και κάποιες από τις ανησυχίες που έχουμε μετά από τα συζήτηση που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Καταρχάς, εάν ακολουθήσουμε την άγουσα της ε, επιβολής κυρώσεων στις, ε, ε, στη βιοενέργεια, να μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι η βασική πηγή ενέργειας, είναι το 60% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης σε ΑΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται ότι θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη των στόχων του 2020 και για, ε, για τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια του 2030. Ε, αυστηρά κριτήρια λοιπόν μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την ικανότητα των κρατών μελών της Ένωσης όχι μόνο να επιτύχουν τουλάχιστον 27% στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και τους υψηλότερους στόχους που προτείνει το Κοινοβούλιο. Ακούσαμε 30-45% μέχρι τόσο φτάσαμε. Δεύτερον, όσον αφορά τη βιομάζα από τα δάση, ελοχεύει ο κίνδυνος αν αποκλείσουμε κάποιες ζωοτροφές από δασική βιομάζα, ε, και το οποίο κατά την άποψή μας ε, δεν δικαιολογείται ε, από τεχνική σκοπιάς και επίσης δεν ξέρουμε και κατά πόσον επιτυγχάνεται από τεχνική σκοπιάς. Ε, διότι θα πρέπει να περιληφθεί αυτό και στο στόχο της βιώσιμης διαχείρισης των δασών. Τρίτον, η εφαρμογή του κριτηρίου βιωσιμότητας και για πολύ μικρής κλίμακας ε, εγκαταστάσεις θέρμανσης. Ο εισηγητής εδώ προτείνει 1 ε, μεγαβάτ ε, όριο. Κατά την άποψή μας, δεν είναι αναλογικό γιατί οι βελτιώσεις που προκύπτουν για το περιβάλλον δεν αντισταθμίζουν το πολύ υψηλότερο διοικητικό κόστος. Επίσης, 85% απέτηση απόδοσης για τη βιοενέργεια ε, και εγκαταστάσεις ε, CHP ε, σημαίνει ότι όλη η βιομάζα και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αυτήν δεν θα είναι βιώσιμη. Κατά την άποψή μας, μόνο κάποιες εγκαταστάσεις στη Σουηδία μπορούν να επιτύχουν αυτό το στόχο. Τέλος, η εφαρμογή ενός ορίου 70% ε, για εξοικονόμηση εκπομπών και ε, για ε, συγκεκριμένους συντελεστές σε όλα τα εργοστάσια βιομάζας ουσιαστικά θα εξαφανίσουν όλα τα συμβατικά βιοκαύσιμα που βασίζονται σε καλλιέργειες μέχρι το 2020. Η πρόταση λοιπόν ουσιαστικά θα έχει τα αποτελέσματα πολύ νωρίτερα από όσο προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, παρά το γεγονός ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από την Επιτροπή για τη μείωση των βιοκανσίμων. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Άικχαλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τις ε, παρεμβάσεις τους και την καλή συζήτηση. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πιστεύω ότι πολλούς ε, από τους στόχους τους έχουμε κοινού και πιστεύω ότι αυτό είναι θετικό. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια μόνο για το θέμα συγκεκριμένα του περίφημου παρατήματος 9, ε, το οποίο ανέφεραν και πάρα πολλοί συνάδελφοι, κ. Λάινεν για παράδειγμα και ο συνάδελφος κ. Χάιτομα, ο οποίος είχε τον τεζαβού του. Πρέπει να το εξετάσουμε, γιατί θεωρώ ότι και εγώ εκ πρώτης όψεως δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει το παράρτημα 9 και συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Χάιτουμα εξ ονόματος του Νίλσα. Πρόκειται για να είναι πραγματικά πολύ μη ευέλικτο τρόπο πρόθεση των ΑΠΕ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει περιθώριο για τα νέα προϊόντα τα οποία μπορεί να εισέλθουν στην αγορά και όταν προωθούμε κάποιες εφαρμογές για τις οποίες γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικέ βιομηχανικές εφαρμογές πρέπει να ξέρουμε και να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση στο σημείο αυτό και γι' αυτό προτείνω το θέμα των έμεσων εκπομπών προκειμένου να ληφθεί υπόψη ακριβώ το στοιχείο αυτό. Παρεπιπτόντως, θα ήθελα να το τονίσω αυτό γιατί σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για τις σε εκπομπές. Αυτό που εννοώ είναι να ισχύουν μόνο για τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Διαβάζοντας την έκθεση, ενδεχομένως να θεωρείτε ότι αυτό θα ισχύει και όλους τους αφαιρούς σκοπούς. Όχι. Τα κριτήρια των έμεσων εκπομπών θα πρέπει να είναι σαφές ότι αφορούν μόνο τα προηγούμενα βιοκαυσίματα όπου έχουμε καύσιμα όπου έχουμε αυτού του στόχου και ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλε εφαρμογέ. Και πάρε μιλάω για τη μελάσα, μιλάω για τι ζωοτροφέ προ άλλου σκοπού και θα πρέπει να, έχουμε υπόψη, να το έχουμε υπόψη αυτό όταν ζητούμε περαιτέρω εφαρμογέ για το ILOC. Καταλαβαίνω γιατί σα ε, θυμίζει κάτι από το παρελθόν αυτό, αλλά να σα πω ότι έχουμε πει μέχρι το 2030 έχουμε θέσει του στόχου και ελπίζω αυτή τη φορά να τα πετύχουμε καλά χωρίς να ορίσουμε σχετικά κριτήρια, δεν θα γίνει οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των υφιστάμενων καρπόνα για τρόφιμα, γιατί έχει πει για παράδειγμα το Κοινοβούλιο ότι θέλουμε να σταματήσουμε με το φινικέλα για βιοκαύσιμα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να το πετύχουμε αυτό και το άλλο είναι ένας τρόπος προς τον συνάδελφο του ECR να πω ότι δεν θα υπάρξει πλέον ε, καύση απορριμμάτων μετά το 2020. Όχι, δεν είπα αυτό, δεν είπα ότι δεν θα υπάρχει. Είπα ότι δεν θέλω να υπάρχει οικονομική υποστήριξη για την καύση των λιμάτων και αποβλήτων, γιατί πρόκειται για έναν από τους λιγότερο αποτελεσματικούς τρόπους προώθησης και μάλλον μεταχείρισης των καυσίμων, των ε, αποβλήτων. Θα πρέπει να φροντίσουμε την κυκλική οικονομία με σωστό τρόπο, αυτό που λέω απλά είναι ότι η οικονομική υποστήριξη για την καύση των αποβλήτων να σταματήσει, γιατί δημιουργεί μη ανταγωνιστικού όρου. Και κάτι άλλο. Οι ροέ αποβλήτων είναι σημαντικέ. Μιλάμε για 50% που προέρχεται από την δασοκομεία. Άρα, όταν μιλάμε για ροή αποβλήτων, μιλάμε και για την νοσοκομεία σε ό,τι αφορά αυτά που είπε η συνάδελφος από τη Φιλανδία, από την Άλτε. Το γνωρίζω ότι υπάρχει αυτός ο στόχος και δεν θα πρέπει να είμαστε αντίθετοι προς αυτόν, αλλά αυτό μπορούμε να το κοιτάξουμε από κοινού προκειμένου να φροντίσουμε να λυθεί το θέμα σε ό,τι αφορά στον τομέα της δοσοκομείας. Να σας πω ότι τα φιλανδικά μέσα και τα φιλανδικά λόμπι είναι άτεγκτα. Σας προειδοποιώ ότι διαβάζω το φιλανδικό τύπο. Αν από τη μία φωνάζουμε στα φιλανδικό τύπο και από την άλλη θέλετε να συνομιλήσετε μαζί μου, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι ενδεχομένω ε, ότι έχουμε διαφορετικά συμφέροντα. Δεν ξέρω αν προκαλώ εμπρικότητα σε κάποιους τα πίσω καθίσματα. Και τέλος, σε ό,τι αφορά το συνολικό στόχο. Αυτό είναι βασικό. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε για την υλοποίηση των στόχων του Παρισιού, μιλάμε για μία σχεδόν ε, μια οικονομία σχεδόν χωρίς ε, άνθρακα μέχρι τα μέσα του αιώνα. Αν υπάρχει ένα τομέα ο οποίο μπορεί να, να κινηθεί πιο γρήγορα από τη μεταφορά σε, από τη γεωργία, είναι το μέσο της ενέργειας. Και εδώ βασικό σκέλος είναι οι ανανεώσιμες. Ο τομέας λοιπόν της ενέργειας θα πρέπει να, έχει, να μην έχει καθόλου άνθρακα, 0% μέχρι το 2040. Αυτό συνεπάγεται το Παρίσι. Άρα το να μιλάμε για το 30% των νεώσιμων μέχρι το 2003 δεν συνεπάγεται εφαρμογή, υλοποίηση των όσων συμφωνήθηκαν στο Παρίσι. Θα πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν καλύτερα αν πραγματικά έχουμε πάρει το Παρίσι στα σοβαρά και θα σας δείξω μέρες, αν θέλετε που καταδεικνύουν ότι ο στόχος του Παρισιού ουσιαστικά συνεπάγεται 45%. Τώρα μάλλον ολοκληρώθηκε και ο χρόνος που είχα για να μιλήσω. Θα σταματήσω λοιπόν και προσβλέπω στη συνεργασία με τους σκιώδεις για να βρούμε συμβαστικές προτάσεις. Σας ευχαριστώ. Για το χρονοδιάγραμμα, 5 Ιουλίου είναι η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Στην Επιτροπή του Περιβάλλοντος η ψηφοφορία θα λάβει χώρα κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε στο επόμενο θέμα εφαρμογή της μακροπεριφερειακής στρατηγικής η κυρία Μίρια Μποζόν είναι η συγγήτρια και θα τη δώσω πάρα αυτό το λόγο. Eh, eh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε από τη συνάδελφη. Δυστυχώ θα χρειαστεί να φύγω πριν το τέλος της συζήτησή μα γιατί έχω την πτήση μου που πρέπει να προλάβω. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιότητες συζητητές για την ε, συνεργασία και τους συναδέλφους. Το 2009 με την απόφαση του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, έδωσε την δυνατότητα να δημιουργηθεί μια στρατηγική για την Βαλτική μετά το 2011 είχαμε μια γενική περιφερειακή στρατηγική για την περιοχή των Άλπων και μετά για την Αδριατική. Έχουμε σήμερα πλέον τέσσερις μακροπεριφέρειες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 19 κράτη-μέλη της Ένωσης και επίσης χώρες που ε, δεν είναι μέλη της ε, Ένωσης. Μέσω αυτών των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών για την επίλυση προβλημάτων που κάθε ένα κράτος ε, μόνο του δεν θα μπορούσε να επιλύσει. Έχουμε δηλαδή μια διακυβερνητική προσέγγιση στα διάφορα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αξιολογεί τις ε, εξελίξεις και κάνει μια έκθεση κάθε δύο χρόνια. στην οποία συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις. Κάθε μια από αυτέ τι τέσσερι μακροπεριφερειακέ στρατηγικέ, βέβαια, έχει τι δικέ τη ιδιαιτερότητε. Ε, το 2016 είχαμε την πρώτη έκθεση τη Επιτροπή, η Επιτροπή Περιφερειακής ε, έκανε μια δική της έκθεση ίδιας πρωτοβουλία. Και χρησιμοποίησαμε ε, εμείς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτής της ε, έκθεσης που είναι πολύ χρήσιμα ιδίω όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι μπορούμε να μετρήσουμε ε, την πρόοδο που σημειώνεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Για να γίνεται αυτό χρειάζεται να έχουμε αξιόπιστους δείκτες ε, στην Αδριατική και στο Ιόνιο ε, το σημαντικό ζήτημα στο οποίο στέκεται η μακροπεριφερειακή στρατηγική από την πλευρά του περιβάλλοντος είναι τα απορρίμματα στη θάλασσα και ε, η γεωργία. Οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτήν προσπαθούν από κοινού να αντιμετωπίσουν τα οικολογικά προβλήματα που σχετίζονται με αυτά. Στο Δούναβι το ζήτημα ήταν οι πλημμύρες που προφανώς δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα στις χώρες που, ε, από τις οποίες διέρχεται ο Δούναβης. Και εδώ προσπαθούμε, προσπαθούν να συνεργαστούν οι χώρες αυτές για την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Τα ευρωπαϊκά ταμεία και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής κατά την άποψή μου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εδώ. Τα καλύτερα αποτελέσματα την έχουμε στη μακροπεριφερειακή στρατηγική Βαλτικής. Ε, όμως εδώ ε, θα έπρεπε να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στην, στα ζητήματα του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα ε, στα ζητήματα της μόλυνσης και της θάλασσας και του, του, του γλυκών νερών και της ατμόσφαιρας που είναι μέρη, με, μέρη της στρατηγικής. Εδώ τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν σε αυτή τη μακροπεριφερειακή στρατηγική θα έπρεπε να θέσουν στόχους οικονομικής φύσεως και ε, σχετικούς με την, την ανάπτυξη του τουρισμού τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα σκιώδη συζητητέ από το ΕΛΚ ο κύριο Τόρφων. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και νομίζω ότι η συνάδελφος μπορούσε να μας επέβαλε μια έκθεση με την οποία μπορώ να συμφωνήσω στο μεγαλύτερο βαθμό. Όπως είπε η συνάδελφος, έχουμε τέσσερι μακροπεριφερειακές στρατηγικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μεμονωμένε υποθέσει αυτές οι στρατηγικές. Ε πολλοί πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση α, καλύπτονται από αυτές τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι σωστό να κάτσουμε να σκεφτούμε πώς λειτουργούν και τι πετυχαίνουν τελικά. Και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να κοιτάξουμε τι θετικέ επιπτώσει τη μακροπεριφερειακή πολιτική και για τον πολίτη. Και να καταστεί σαφή ε, ποια είναι η πολιτική αυτή και τι συνέπειε έχει. Γιατί δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνεται αυτό παρατητάω, ο πολίτη. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντική αυτή η έκθεση και πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε πώ την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο θα μπορούσαν αυτέ οι μακροπεριφερειακέ στρατηγικέ να ενσωματωθούν στο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και η βασική σκέψη είναι ότι δεν υπάρχουν ε, ξεχωριστά κονδύλια για την ε, στρατηγική αυτή. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς στα επιστάμενα προγράμματα, στον ορίζοντα, στο κόσμο, ε, Interreg, τα κατά ταμεία, μπορούν να λάβουν ιδιαίτερη σημασία οι μακροπεριφερειακές αυτές τις πολιτικές. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ήδη είπε η συνάδελφος, αλλά στις διάφορες μακροπεριφερειακές στρατηγικές, όταν μιλάμε για βιωσιμότητα, για προστασία του περιβάλλοντος, υπάρχουν ε, πάρα πολλές προκλήσεις, αλλά και πάρα πολλές ευκαιρίες. Εγώ είμαι από τις Άλπες, για παράδειγμα. Και το θέμα της αλλαγής του κλίματος εδώ αποτελεί σίγουρα μεγάλη πρόκληση, αλλά για παράδειγμα το θέμα και το σχέδιο της ε, βιώσιμης μεταφοράς, ε, μεταφορών αποτελεί και μια μεγάλη ευκαιρία προκειμένου αυτός ο χώρος να διαμορφωθεί α, με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμείνει βιώσιμος στη μακροπεριφερειακή πολιτική και κυρίω ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση αυτή τη πολιτική, θεωρώ ότι θα πρέπει να κάτσουμε και να εξετάσουμε συγκεκριμένα τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται. Και αφενός, όπως ακούσαμε, το θέμα είναι πώς θα ενσωματωθούν τα εφιστήμενα ταμεία προκειμένου να συνεχίσουν να υπάρχουν και έχω και παράδειγμα υπόψη μου το Interreg πώς μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στη μακροπεριφερειακή πολιτική και κοιτάξτε, θα, πρέπει να σκεφτούμε γιατί είμαστε στην αρχή της διαδικασίας πώς τα καινούργια ε, χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το ΕΦΣΥ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για έργα βιωσιμότητα στη μακροπεριφερειακή πολιτική και πώς μπορεί να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο το ΕΦΣΥ ώστε να έχουν ιδιαίτερη σημασία και να προτιμούνται τα διασυνοριακά προγράμματα. Αυτό θα ωφελούσε ασφαλώς την μακροπεριφερειακή στρατηγική και θα βοηθούσε ασφαλώς να προωθηθούν τα βιώσιμα αυτά σχέδια και τα περιφερειακά αυτά σχέδια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Κυρία Μέιζερ από την Άλτε. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ε, εξονόματος της κυρίας Μίλλερ θα μιλήσω. Ξέρω, ξέρω ότι με βλέπετε. Σας ευχαριστώ και να ευχαριστήσω και την ε, εισηγήτρια για την έκθεση που αποτελεί καλή βάση για την ε, μελλοντική μας εργασία. Οι μακροπεριφερειακές πολιτικές είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσο για το κλίμα και το περιβάλλον, γιατί τα προβλήματα συνήθως είναι ε, διασυνοριακά και μπορούν να επιληθούν καλύτερα με συντονισμό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δυστυχώς ε, δεν λαμβάνει τόσο υπόψη τις πρακτικές ε, συνέπειες των τεσσάρων αυτών μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Δεν έχει και πολύ χρόνο βέβαια στη διάθεσή της, είναι λογικό. Πολλά λοιπόν θα πρέπει να βελτιωθούν. Οι πρακτικές συνέπειες θα πρέπει να μπουν στο επίκεντρο για τη μελλοντική, το μελλοντικό προσανατολισμό της δημοκρατική ε, πολιτικής. Έχουμε δύο σημεία τα οποία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Καταρχάς, οι προκλήσεις αυτές ε, μόνο μακροπρόθεσμα μπορούν να επιληθούν και αυτό είναι αντίθετο με την ε, προσανατολισμό των έργων για τα κονδύλια. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε σίγουρα τη μακροπρόθεσμη διάσταση όταν αφορά τη χρηματοδότηση των μέσων αυτών. Κατά δεύτερον, η πρακτική εφαρμογή τέτοιων έργων μπορεί να σημειώσει επιτυχία αν τα μέτρα αυτά γίνουν αποδεκτά και από τους ντόπιου. Αυτό τι σημαίνει ότι χρειάζεται απαραίτητα διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης, τα μέτρα θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η πεθρός αποτελεί και ένα τρόπο ζωής και μπορεί να θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει συντονισμός με τον τρόπο αυτό που δουλεύουμε και που ασκούμε την οικονομική δραστηριότητα. Ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, θα ήθελα να δώσω τον ε, λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε θα ήθελα εκ μέρους της Επιτροπής να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής για την πολύ ισορροπημένη ε, πρόταση, το πολύ ισορροπημένο σχέδιο έκθεσης και την εισηγήτρια βεβαίω ευχαριστούμε. Την υποστηρίζουμε. Μια παρατήρηση σε σχέση με την τελευταία παρέμβαση. Είναι απόλυτα σωστό το γεγονός ότι η έκθεση ε, τη επιτροπή δεν καταλήγει σε συμπεράσματα σε κάποια θέματα, διότι θέλαμε να ξεκινήσουμε και κάπω τη συζήτηση. Θα δείτε ότι στα συμπεράσματα έχουμε τρει ερωτήσει που θέτουμε στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και στα άλλα θεσμικά όργανα για να ξεκινήσει η συζήτηση για τα θέματα αυτά όσον αφορά τις προτάσεις στο σχέδιο γνωμοδότησης, όπως ε, σας είπα, ε, πολύ που μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Μία μικρή παρατήρηση ίσονο σημασία. Στο σημείο 7 αναφέρεται το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τομέας αυτός για την προσαρμογή, ίσως θα έπρεπε να αναφέρεται ο όρος adaptation, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ε, κατά τα λοιπά, θεωρώ ότι είναι πολύ ισορροπημένη πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. 6 Ιουλίου, 11 η ώρα, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Ψηφίζουμε 28 Φεβρουαρίου, ε, Σεπτεμβρίου. Συγγνώμη. Η Ρέτζη θα ψηφίσει 9 ή 10 Οκτωβρίου και ε, ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο κατά πάσα πιθανότητα. Αυτά λοιπόν για το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης και τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης να ενημερώσω τα δύο μέλη που έχουν την καλοσύνη να μείνουν εδώ μαζί μας, πέρασε και η ώρα, ότι οι επόμενες συνεδριάσεις θα γίνουν 10, 11 ε, και 12 Ιουλίου στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και καλή σας μέρα.